Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτη ψηφοφορία για το σημείο 13 ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρίφαλου. Έχουμε μία ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται. No. Everybody voted. The vote is closed. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Όχι, συγγνώμη. Ναι, αφού ψήφισε και ο Τζο μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο είναι το... Το σημείο 14. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 για την έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου BT11 κτλ. Και γι' αυτό θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody had voted. Ψηφίσατε όλοι. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Now we can go to the next item in our agenda. Προχωράμε στο επόμενο θέμα της της διάταξης, αφού ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Ετήσια έκθεση 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Έχουμε μία γνωμοδότηση και η συγγητής μας είναι η, συνα... Συνάδελφοι, πριν να ξεκινήσουμε, Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί βοηθοί, Άξελ. To continue to speak, is a lot Εάν θέλεις να συνεχίσεις να μιλάς, έχει χώρο απ' έξω από την αίθουσα. Για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε την εργασία μας εδώ. Το λόγο έχει συνάδελφος Ντογνανό, που είναι η συγγήτρια για την γνωμοδότηση. Η κυρία Ντογνανό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας παρουσιάζω αυτή την ε, γνωμοδότηση, ε, διότι αυτές οι αρχές βρίσκονται στα θεμέλια της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού δομήματος. Ε, ο στόχος είναι να ε, δώσουμε σάρκα και ωστά σε μια ε, απόφαση που έχει ληφθεί ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό να ξεφύγουμε από, την, το απλό γράμμα της ε, ε, πρότασης Κομισιόν ε, και να σχολιάσουμε την πρόταση αυτή. Δύο ιδέες χαρακτηρίζουν την νομοδότησή μου. Πρώτον, διαπιστώνουμε ότι τη σημασία αυτών των αρχών για τις πολιτικές ε, οι οποίες απασχολούν την Επιτροπή μας. Και δεύτερον, σημασία της εμπιστοσύνη στην μεταβίβαση της κυριαρχίας ε, που συμβαίνει όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ένα πιο ευρύ κύκλο και ε, σε πιο μακρινό επίπεδο. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην σημασία ότι η ε, Επιτροπή μας όταν ελέγχει την αναλογικότητα και την επικορικότητα πρέπει να ισορροπεί την, τα τρία επίπεδα ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό στην εφαρμογή. Το διακύβευμα ξεπερνάει τις χώρες, ε, αλλά ταυτόχρονα ε, είναι και εθνικό και τοπικό. Και αυτά θα πρέπει να ισορροπήσουμε. Η Επιτροπή έμβει στην κλιματική αλλαγή, στη βιοπικιλότητα, στην ε, ε, διατήρηση της ποικιλομορφίας, ε, ε, χρειάζεται να ληφθούν δράσεις σε υπερεθνικό επίπεδο. Η απόφαση, η παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγγυώνται μια αποτελεσματική πολιτική διότι το διακύβευμα όπως είπαμε πολλές φορές ξεπερνάει το εθνικό πλαίσιο. Γι' αυτό το λόγο υπογραμμίζω τη σημασία της Επιτροπής μας στην ε, στο σχεδιασμό και την επεξεργασία και σε τεχνικό επίπεδο των προτάσεων. Και βασίζομαι στην, ε, στο γεγονός ότι επί των πέντε προτάσεων της ε, Κομισιόν που έλαβαν τις πιο πολλές αιτιολογημένες γνώμες το 2014, δύο από αυτές τις πέντε δύο εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Οπότε υπάρχει θέμα επικορικότητας και αναλογικότητας σε μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν την Επιτροπή μας πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Ο έλεγχος της επικορικότητας και της αναλογικότητας ε, δίνει ένα δυναμισμό ε, στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγυάται την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους. Το να εξασφαλίσουμε την, τον καλύτερο σεβασμό αυτών των αρχών ε, σημαίνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε πως αυτά τα θέματα πολλές φορές επίμαχα θα ε, υλοποιηθούν με τρόπο αποτελεσματικό, ρεαλιστικό ε, και αυτό θα ωφελήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της στο μέλλον. Τα απόβλητα και η κυκλική οικονομία ή ε, τρόποι για να ε, ε, ε, σε τέτοιου θέματα ο τρόπος να πετύχουμε τους στόχους μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός κάθε φορά. Θα πρέπει λοιπόν να ε, συντονίσουμε ακόμα περισσότερο τις πολιτικές μας. Οι περισσότερες ιδεολογημένες γνώμες για την πρόταση σχετικά με τα απόβλητα αμφισβητούσαν την, ε, το ρεαλισμό των στόχων, την αδυναμία να, πετύχ, τους πετύχουμε ή την το γεγονό ότι οι πρόσθετοι στόχοι αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών ε, μελών ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε κράτου μέλου. Χρειάζεται λοιπόν ρεαλισμό και αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε ενισχυμένη αναλογικότητα και επικουρικότητα. Ένας ρεαλισμό λοιπόν και μια αποσαφήνιση των στόχων μέσω πρόθεσμα ε, και έλεγχο των προσπαθειών που έχουν ήδη γίνει. Οι προσπάθειε έχουν ήδη γίνει, αυτό το ε, έχουν κάνει οι πολλοί συνάδελφοι όπως για παράδειγμα στις εκπομπές ε, ρήπων ε, ένα επιχείρημα το οποίο θα το ξαναδούμε συχνά στο μέλλον. Ο κίνδυνος να βγούμε από τις, να, να μη συμμορφωθούμε με τις αρχές επικοινωνικότητα και της αναλογικότητας είναι μεγάλος και γι αυτό, λόγο, γι' αυτό λόγο θα πρέπει να το αποφύγουμε προκειμένου να αποφύγουμε και καθυστερήσεις στην επεξεργασία των προτάσεων. Επίσης, θα ήθελα αργότερα να υπογραμμίσω το εξής. Η αποδοχή της ε, μεταφοράς της κυριαρχίας ε, ε, πρέπει να συνοδεύεται από εμπιστοσύνη στα όργανα που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική η ανάγκη ελέγχου και διαφάνειας των ε, κοινοτικών υπηρεσιών και οργανισμών, των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μεγάλη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποιοι θα εκπλαγούν από αυτό που θα πω, αλλά το θέμα πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί. Ε, το να δεχτούμε την εκχώρηση κυριαρχίας έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με θεμητό τρόπο σε ανώτερο επίπεδο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε εγγύσεις ε, ότι η πολιτική αυτή σε ανώτερο επίπεδο θα υλοποιείται ε, με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό έχει σχέση με την επικουρικότητα. Το θέμα είναι αν πράγματι αυτό το ανώτερο επίπεδο είναι ε, αποτελεσματικό. Όμως το, ε, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση 15 του 2012 λέει ότι οι συγκρούσει συμφερόντων δεν τη επαρκού επαρκούς διαχείρισης εντός της ΕΦΣΑ. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις της ΕΦΣΑ δεν είναι απαραίτητα άψογες. Τελο πάντων δημιουργούνται αμφιβολίες. Η εκχώρηση κυριαρχίας λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι θεμητή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι λοιπόν ένας άλλος τρόπος να δούμε την ε, επικορικότητα ε, με βάση όχι μόνο την, ε, ε, το νομοθετικό έργο. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω τελειώνοντας και το εξής. Αυτή η διαδικασία ε, σχεδιασμού της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, θα πρέπει να δώσει περισσότερα, ε, ισχυρότερο ρόλο στα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου να ενισχυθεί η αρχή της αναλογικότητας και της, απο, της Αυτό συνδέεται με το προηγούμενο επιχείρημά μου, διότι βλέπουμε πως η επικουρικότητα και η αναλογικότητα είναι στόχοι, δυναμικοί στόχοι και κανόνες. Σε αυτή την κατακόρυφη σχέση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το καθοδικό ρεύμα. Το πώς δηλαδή εφαρμόζονται οι, ε, τα, νομο, τα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα το ανωδικό ρεύμα, το πώς δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να βοηθήσουν στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πράσινη κάρτα για παράδειγμα ε, που προτάθηκε από ορισμένα κοινοβούλια είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε διότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε την θετική συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το επιχείρημα είναι παρόμοιο και σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα ε, εργαλείων εφαρμογής. Είναι πιθανό μερικές φορές οι προτάση της ε, Κομισιόν ε, να χρειαστεί να προσαρμοστεί. Οι προτάσεις της Κομισιόν να χρειάζεται να προσαρμοστούν Αυτά ήθελα να πω. Ε, δεν ήθελα απλώς να σχολιάσω την έκθεση της Κομισιόν. Προτείνω μια επικοδομητική κριτική. Είναι καθήκον μας να δρούμε προς όφελος των ε, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά και ε, εγκύτερα στους Ευρωπαίους πολίτες. Περιμένω τα σχόλιά σας, τα σχόλια των συναδέλφων μου, σε συνεργασία με τους οποίους και συμβιβαστικά θα ενισχύσουμε το σκελετό της έκθεσης τον οποίο σας παρουσίασα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει ο πρώτος γύρος των σκιωδών εισηγητών. Η κυρία Γκαρτίνη, εξ του κυρίου Πατριτσέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διαβάζω την παρέμβαση που είχε προετοιμάσει ο συνάδελφος Πατριτσέλο που αρχίζει βεβαίως ευχαριστώντας ε, στο όνομα της πολιτικής ομάδας ε, του ΕΛΚ την εισηγήτρια Ντορνανό για την εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα για τα θέματα ε, της αναλογικότητας και της επικουρικότητας που είναι βασικές αξίες, αρχές για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Όπως ορίζεται από το άρθρο 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας στους τομείς που δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διπλή ε, λειτουργία. Από τη μια πλευρά έχουμε την αρχή που επιτρέπει την επισκόπηση τη δυνατότητα λήψη αποφάσεων των κρατών μελών στην περίπτωση που ένα θέμα μπορεί να ρυθμιστεί με αποτελεσματικό τρόπο σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από την άλλη πλευρά είναι καλό να θυμίσουμε ότι η ίδια αρχή νομιμοποιεί την παρέμβαση της Ένωσης όταν τα κατημέλη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν ε, στόχους που έχουν οριστεί με ικανοποιητικό τρόπο, σε ικανοποιητικό βαθμό και άρα η ευρωπαϊκή παρέμβαση μπορεί να επιφέρει μια σημαντική προσθέμενη αξία. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει περαιτέρω ενισχύσει την αρχή της επικουρικότητας, θεσπίζοντας διάφορους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να επαληθεύεται η σωστή συμμόρφωση προς τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας. Μεταξύ αυτών οι αιτιολογημένες νομοδοτήσεις που αποτελούν το μέσο δια του οποίου τα εθνικά κοινοβούλια μέσω αναδρομικών αξιολογήσεων καθορίζουν κατά πόσο οι δράσεις που έχουν υιοθετηθεί σε κοινοτικό επίπεδο είναι κατάλληλα, συνεπείς, αποτελεσματικές Σκόπιμε και περιέχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ω προ αυτό λοιπόν, όσον αφορά την ετήσια έκθεση 2014 για τα θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας, έχει καταγραφεί σημαντική μείωση των αιτιολογημένων νομοδοτήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, αυτή η μείωση οφείλεται στη σημαντική μείωση της ε, συνόλου των νομοθετικών προτάσεων που έχει οθετήσει ε, η Κομισιόν στην τελική φάση της εντολής της και άρα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ένα μήνυμα μικρότερου δείγμα μικρότερου ενδιαφέροντος σε σχέση με τα εθνικά ε, κοινοβούλια, από πλευρά μάλλον των εθνικών κοινοβουλίων για την επικουρικότητα, ε, ε, χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βελτιώνοντας τον πολιτικό διάλογο σε διάφορα, στα διάφορα επίπεδα τα θεσμικά και ενισχύοντας τις δυνατότητες των εθνικών κοινοβουλίων να εκφράσουν γνωμοδο, γνώμες, γνωμοδοτήσεις για τα σχέδια των ε, τα κοινοτικά σχέδια. Ο πολιτικό διάλογο ανάμεσα στη Κομισιόν και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει έχει εντατικοποιηθεί και χάρη στι διάφορε επισκέψει των Επιτρόπων στι ε, εθνικέ νομοθετικέ συνελεύσεις ώστε να αναλύσουν και να παρουσιάσουν τα προγράμματα και τι νομοθετικέ προτάσει ω πολιτική ομάδα λοιπόν για αυτού του λόγου θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση πεπισμένη όπω στηρίζει και η πρόσφατη διαθεσμική ε, ε, συμφωνία που έγινε την προηγούμενη το προηγούμενο Σεπτέμβριο ανάμεσα στα ε, Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα μόνο αν οι θεσμοί μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σε με σεβασμό των διαδικασιών που προβλέπουν οι συνθήκες θα συνεχίσουν να τηρούν αυστηρά τις βασικές αρχές του ε, ε, κοινοτικού δικαίου, δηλαδή την δημοκρατική νομιμότητα, την επικουρικότητα, την αλογικότητα και τη βεβαιότητα του δικαίου. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, συνάδελφος, αντικαθιστώντας τον κύριο Τζεντήλε, ο κύριος Καπούτο. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο τον άνο για την εξαιρετική της εργασία οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας είναι κατευθυντήριες αρχές της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, της ορθής, και η ορθή τους αξιολόγηση εξαρτάται από την εγκυρότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ε, πολιτικών. Θετικό στοιχείο είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή τα τελευταία χρόνια των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διαδικασία, αλλά απόρροπα έχουμε ακόμα από την πλήρη του εμπλοκή. Οι περισσότερε γνωμοδοτήσει των Εθνικών Κοινοβουλίων, ακόμα και για θέματα περιβάλλοντο, προέρχεται από λίγα κρατημέλη και γι' αυτό τα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να τοποθετήσουν τα ευρωπαϊκά να, να διευκολύνουν τα, τα εθνικά κοινοβούλια να ελέγξουν τις νομοθετικές προτάσεις ε, και να τους παρέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις για τις αποφάσεις τους μέσα στο πλαίσιο, μάλλον, όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Είναι απαραίτητο τα εθνικά κοινοβούλια να εκδίδουν ε, αιτιολογημένες νομοδοτήσεις, όχι μόνο για τα νομοθετικά ε, κείμενα της Επιτροπής, αλλά και για τα μη νομοθετικά κείμενα που προηγούνται τις διαδικασίες ε, νομοθέτησης, ώστε να αιτιολογηθούν καλύτερα οι μελλοντικέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε τη Ένωση. Θεωρώ πω είναι απαραίτητη η υιοθέτηση κοινών προτύπων, επί τη βάση των οποίων τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούν να παρέμβουν, γιατί οι αιτιολογημένε νομοδοτήσει, έτσι όπω παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, δεν ε, είναι πάντοτε χρήσιμες γιατί διαφέρουν ε, λόγω της μορφής και το είδος της επιχειρηματολογίας τους. Ευχαριστώ πολύ. με Μέκερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντόχναγνου για τη δουλειά της. Είναι μια πολύ καλή αρχή. Η δική μας πολιτική ομάδα ECR εδώ και χρόνια πρωτοστατεί ε, στην προσπάθεια για καλύτερη νομοθεσία η Αναλή Βανμποσόιτ που είναι και από το ίδιο μου το κόμμα και την αντιπροσωπεία ασχολείται με αυτά. Οι κανόνες θα πρέπει να ενθαρρύνουν και όχι να αποθαρρύνουν και να απογοητεύουν. Θα πρέπει να αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κρίσιμο για να επανέλθει αξιοπιστία των Ευρωπαίων πολιτών. Η αρχή της επικορικότητας και της αναλογικότητας είναι αρχές βασικές και σημαντικές για την ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία και την περιβαλλοντική. Τα θέματα του περιβάλλοντος ε, καλύπτουν ένα τομέα που είναι συντρέχουσες οι αρμοδιότητες. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η βιοπικιλότητα, η κυκλική οικονομία, το κλίμα, όλα αυτά είναι διασυνοριακά, άρα και οι λύσεις θα πρέπει να είναι διασυνοριακές. Είναι λοιπόν ένα τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει και οφείλει να δείξει τη θέμενη αξία, την αξία της. Τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, η συγκήτρια τονίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην εκτέλεση και υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Υπάρχουν όμως κράτη-μέλη, όπως το δικό μου, το Βέλγιο, όπου πάει παραπέρα αυτό. Οι περιφερειακές διοικήσεις, όπως είναι η Φλάνδρα, η περιφέρεια που εγώ εκπροσωπώ, έχουν πλήρες αρμοδιότητες και εξουσίες και κυριαρχία και θα παρακαλούσα να το γράφει και το κείμενο αυτό. Δεύτερον, έχει σχέση με το προηγούμενο. Η κατανομή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων οδήγησε στο εξή. Τα περιφερειακά κοινοβούλια έχουν συνυπευθυνότητα για την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου επί των ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο Βέλγιο είναι και μοναδική η κατάσταση, διότι μεταξύ των κοινοβουλίων που έχουμε Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και Περιφερειακά, δεν υπάρχει ιεραρχία ε, και τα δύο θεωρούνται ισότιμα εθνικά κοινοβούλια. Στη συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζεται αυτό επίσης ε, και παίζουν από κοινού ένα σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται για ε, την εποπτεία, ε, για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Γι' αυτό έχει σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά να λάβει υπόψη της ότι σε κάθε κράτος μέλος μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Και εμάς λοιπόν το Κοινοβούλιο μας θεωρείται εθνικό το περιφερειακό. Και τρίτον, προτείνεται για μια, μια διαδικασία πράσινης κάρτας πρέπει να τολμήσουμε, αν το συζητάμε αυτό, να συζητάμε και μια α, διαδικασία κόκκινης κάρτας. Θα πρέπει δηλαδή να πίπτει και ράβδος καμιά φορά και να μπορούν ε, τα ε, κοινοβούλια, τα εθνικά στο βαθμό που τους αναλογεί, να ε, απορρίπτουν και να επιστρέφουν νομοθεσία. Γιατί το δημοκρατικό έλλειμμα καλύπτεται από ε, ελέγχους από τα εφιστάμενα όργανα και όχι με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους. Προς το παρόν, λοιπόν, ε, σταματώ εδώ και θα κάνω και σχετικά τροπολογίες για όλα αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ φυσικά πρώτα απ' όλα την κυρία Ντοχνανό Γιατί ο έργο θα είμαι πολύ σύντομος. Ακούσαμε ήδη τα κυριότερα σήμερα. Δεν πρέπει να κάνουμε αφηρημένες πολιτικές συζητήσεις για τους γενικούς κανόνες της επικουρικότητας και της ε, αναλογικότητας και να αφήσουμε εκτός του πεδίου όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας, την ε, Επιτροπή Ένβη. Δεν είναι σκόπιμο να κάνουμε αφηρημένες συζητήσεις, ούτε είναι καλός τρόπος ε, εργασίας αυτός. Θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τα θέματα που αφορούν τη δική μας επιτροπή σε αυτό το ε, κείμενο, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Γιατί εδώ συζητάμε γενικά όπου υπάρχει μια διελκυστίδα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. και των διαφόρων επιτροπών για την επικουρικότητα και ποιος αποφασίσει τι πράγμα. Αυτό λέγεται και επιτροπολογία. Θα μπορούσαμε ίσως να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση αυτή, τονίζοντας πολύ ειδικά θέματα που αφορούν τη δική μας Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επίσης θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση αυτή βλέποντας και πέρα από το 2014. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία, τη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα κτλ. Μπαίνουμε σε θέματα πάρα πολύ ουσιαστικά και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Αυτά για σήμερα προς το παρόν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Η κυρία Μινέρ. Όχι, δεν είναι εδώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνώ με τον Νίλς ότι δεν θα πρέπει να μπούμε σε μια γενική συζήτηση περί της αναλογικότητας και της επικορικότητας. Αυτό μπορεί να γίνει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, και όποιο ενδιαφέρεται ας πάει εκεί, ήδη η συζήτηση αυτή λαμβάνει χώρα εδώ και πολύ ώρα. Εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε στις περιβαλλοντικές πτυχές. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Μέρσμάκερ ότι οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δίνουν προστιθέμενη αξία. Και ε, όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την ασφάλεια των προϊόντων, δημόσια υγεία κλπ. Εκεί ακριβώς είναι σημαντική η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μέχρι τώρα η, η διαδικασία της επικορικότητας χρησιμοποιεί το αρνητικά για να μπλοκάρει κάτι, να το φρενάρει. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια ότι υπάρχει και μια θετική προσέγγιση της επικορικότητας. Όταν θεωρούμε ότι η Κομισιόν ε, αμελή να λάβει δράση. Ακόμα και αν ένα περιφερειακό κοινοβούλιο το θεωρεί, θα πρέπει αυτό για να βοηθήσει τους βέλους συναδέλφου. θα πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία. Ε, ο κύριος ε, Κάμερον για την κόκκινη κάρτα κάτι έχει ήδη κάνει. Δεν, είστε το, δεν είναι το πολιτικό σας αφεντικό, εντάξει. Νόμιζα ότι ήταν από την ομάδα σας. Νομίζω ότι ο κύριος Κάμερον ήδη έχει αναλάβει δράση για το θέμα της κόκκινης κάρτας με τη συμφωνία για το Brexit. Ε, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι για την επικορικότητα θα πρέπει ε, να ξεπεράσουμε το ποιο είναι το πιο καλό επίπεδο λήψη των αποφάσεων. Ε, πολύ συχνά ξεπερνάμε την κίτρινη κάρτα, τη διαδικασία κίτρινη κάρτα. Ε, γιατί ο κόσμο αρχίζει και χρησιμοποιεί την επικορικότητα για να μπλοκάρει κάποιο νομοθέτημα το οποίο δεν του αρέσει το περιεχόμενό του. Η, το τεστ τη επικορικότητα δεν αφορά αυτό. Αφορά το κατά πόσον οι αποφάσει λαμβάνονται στο ορθό επίπεδο. Και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πολύ συχνά επικρατεί σύγχυση. Κάποιοι που δεν του αρέσει ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα λένε βγάζω κίτρινη κάρτα. Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Αν δεν αρέσει κάποιον μπορεί να τροποποιηθεί ενδεχομένως, αλλά η επικουρικότητα δεν αφορά αυτό. Και σε θέματα εσωτερικής αγοράς σας είμαστε ειλικρινείς. Ε, πολύ συχνά χρειάζεται να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια προϊόντων. Για παράδειγμα το REACH, ε, τα νανοηλικά, όλα αυτά μπαίνουν στην αν όλα αυτά μπουν στην ομπρέλα της, ε, του νομοθετήν καλύτερα ε, είναι μια λανθασμένη προσέγγιση η οποία ενδεχομένω προέρχεται από πιέσεις και από λόμπι συγκεκριμένων εταιριών που έχουν ε, συμφέροντα. Μπορεί οι επιχειρήσεις αυτές, οι εταιρείε αυτές να μην θέλουν το συγκεκριμένο νομοθέτημα, το α ή το β νομοθέτημα, αλλά αυτό μπορεί να ωφελήσει τον κόσμο, οπότε θα πρέπει να προχωρήσει και να μην χρησιμοποιείται επικορικότητα για να το σταματήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν ξέρω αν τα απλά μέλη θέλουν το λόγο. Όχι. Η Επιτροπή. Ούτε. Οπότε θα δώσω το λόγο ξανά στην εισηγήτρια, την κυρία Ντορνάνου. Σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω εν συντομία. Κυρία Καρτίνη σε ό,τι αφορά την μείωση των αριθμών των προτάσεων τη Κομισιόν. Σας υπενθυμίζω ότι στο, στην πρώτη παράγραφο της ιδεολογικής έκθεσης θα το δείτε. Ε, βέβαια εσείς λέτε ότι μπορείτε, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα, μπορούμε να αποβάλει τροπο, τροπολογία. Κύριε Καπιτό, η δραστήρια συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, ναι, ε, είναι, ε, καθιστά το σύστημα πιο δυναμικό. Όσο βέβαια πιο λεπτομερείς είναι οι γνωμοδοτήσεις, ε, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η βελτίωση της νομοθεσίας. The Mercy Maker. Ε, η, το ECR, η ομάδα του ECR ήταν πάντοτε επικοδομητική σε αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ για το, τα σχόλιά σας. Μπορούμε να συνεργαστούμε καλά. Ε, μετά, τοπικές και περιφερειακές αρχές και κοινότητες. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ποικιλόμορφη. Συμφωνώ λοιπόν. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί τις ε, τοπικές ιδιομορφίες. Ο κ. Τόρβαλς ε, δεν είναι γενικόλογη η έκθεσή μου, η γνωμοδότησή μου, δεν μπορώ να είμαι όμως πιο λεπτομερής, μια σελίδα έχω. Περιμένω τις ε, τροπολογίες σας έτσι ώστε να γίνει πιο σαφής. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να είστε συγκεκριμένοι. Έτσι ώστε να, στην επόμενη συνεδρίασή μας να διαθέτουμε και συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. 27 Μαΐου. Εδώ θα ψηφίσουμε την 21η Ιουνίου στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Γεωρή Νομικών Θεμάτων στις 8 Νοεμβρίου και το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια με το καλό. Πάμε στο επόμενο θέμα στη Μέση Διάταξη, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέρμανση και την ψήξη. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φιέλνερ για να μας παρουσιάσει το σχέδιο της νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Νομοδότηση σύντομη. Είναι σύντομη και συμπαστική. Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ε, κατανάλωσης ενέργειας ε, είναι, προορίζεται για την ψήξη και τη θέρμανση των κτηρίων. Ε, δεν νομίζω πως είναι κάτι το φυσιολογικό και αυτό είναι το σημείο εκκίνηση. Θέλω να το τονίσω. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας. Και επίσης πολλοί από εμά ε, περάσαμε χρόνο συζητώντας το κίνδυνο μιας κρίσης φυσικού αερίου. Μια τέτοια κρίση θα ήταν και κρίση θέρμανσης. Χωρίς το φυσικό αέριο σήμερα θα ξεπαγιάζαμε. Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή και στην Ένωση είναι το γεγονός ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί. Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες αλλά και περιστάσεις στις διάφορες χώρες. Ισχύουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Διαφέρουμε πολύ όσον αφορά το κλίμα και ε, ε, είναι αδύνατον να βρεθεί χρυσή τομή Υπάρχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι που έχουν διάφορε λύσει να προτείνουν και είναι πολύ καλή, αλλά συνήθω είναι πολύ καλή για ένα μέρο ε, και όχι αλλού. Αυτό που λειτουργεί στην Ισπανία δεν θα λειτουργήσει απαραίτητο και στη Φιλανδία. Ε, γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε ε, στα συστήματα και να έχουμε μία προσέγγιση σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης νομίζω πως χρειάζεται να κρατήσουμε χώρο για να υπάρχει τεχνικώς ουδέτερη προσέγγιση, να μείνει χώρος για την αγορά, ώστε να βρει διαφορετικές λύσεις για τα διαφορετικά μέρη της Ευρώπης. Άλλο παράδειγμα που θέλω να θίξω είναι το γεγονός ότι έχουμε σήμερα, σε αυτή την νομοθεσία που είναι πολύ κατακαιρματισμένη, έχουμε διαφορές νομοθεσίες που στηρίζουν ε, κάποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι όλες. Ε, και αυτό εμποδίζει τη σωστή λειτουργία της αγοράς, ώστε δηλαδή να διευκολυθούν οι προκλήσεις. Ένα από αυτά τα παραδείγματα δε είναι ότι επιτρέπεται να υπολογίσει την, ε, ενέργεια, την παραγωγή ενέργειας, ε, ηλιακής ενέργειας σε ένα σπίτι, αλλά δεν επιτρέπεται να τη λάβεις υπόψη ό, όταν κανείς υπολογίζει την ενεργειακή απόδοση νοστηρίου, να υπολογίσει άλλες ανανεώσιμες που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν παράγονται στο συγκεκριμένο κτίριο. Γι' αυτό και δεν πρέπει πιστεύω να μπούμε στις λεπτομέρειες. Τέτοιου είδους παραδείγματα είναι αυτά που θα πρέπει να δει η Επιτροπή και να τα αντιμετωπίσει. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι σήμερα έχουμε περίπου 25% της ενέργειας για θέρμαση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι παρα, περισσότερο. Και γι' αυτό οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει σε αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να, δηλαδή να στηρίξουμε όλε τι μεθόδου ταυτόχρονα. Και έπειτα πιστεύω επίση, αν και γνωρίζω ότι είναι επίμαχο το θέμα, ότι το θέμα της ενέργεια από τα απόβλητα θα είναι κομμάτι του μείγματο γιατί η κατάσταση είναι πολύ κακή στον τομέα αυτό. Το να είμαστε πολύ σκληροί λοιπόν και να το αγνοήσουμε μπορεί να μας κάνει να μείνουμε στα πολύ άσχημα, πολύ κακά, ορυκτά καύσιμα που θερμανούν τα κτίρια μας σήμερα. Αυτά έχω να πω. Φυσικά περιμένω σχόλια των ε, συναδέλφων, ώστε να γίνει αυτό το κείμενο ε, καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε με τους και οδησίγητες. Ο κύριος Τζόφολη πρώτα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή του εργασία. Εν γέννη ε, τα όσα λέει στην έκθεσή του τα συμμερίζομαι. Όμως υπάρχουν και κάποιες στοιχείες που θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και να βελτιωθούν. Και γι' αυτό είναι η προθεσή μου να υποβάλω κάποιες τροπολογίε. Καταρχάς θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι όπω θυμήσατε στην Ευρώπη η θέρμανση ε, και η ψήξη αποτελούν, καταναλώνουν περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ε, στην Ήπειρο και το 36% εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα οφείλεται στις εκπομπές των δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων είναι λοιπόν τεράστια σημασία για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου, ε, να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να προστατευτεί η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ως προς αυτό θα ήθελα να τονίσω ακόμα ένα στοιχείο, ότι δηλαδή αν από τη μια πλευρά μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο τμήμα των ευρωπαϊκών ε, κτηρίων ε, ε, σπαταλούν ενέργεια λόγω της κακής τους ποιότητας, από την άλλη πλευρά το 11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και είμαστε στο 2016 δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ώστε να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του το χειμώνα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να τεθεί τέλος όσο γίνεται πιο σύντομα σε αυτή την αδικία, εφαρμόζοντας και σε αυτούς τους τομείς της εναρχή της κυκλικής οικονομίας, ε, δίνοντας κίνητρα για παράδειγμα για την παραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού στην, από συμπαραγωγή. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η εμβάθυνση και στο θέμα του district heating. Είναι σημαντική επίσης η πτυχή που πρέπει να αναπτυχθεί, η ενημέρωση του καταναλωτή. Πρέπει δηλαδή ο καταναλωτής να είναι σε θέση να παίρνει πληροφορίες σαφείς και πλήρεις για τα τεχνικά πλονεκτήματα και οικονομικά πλονεκτήματα των νέων εγκαταστάσεων ε, να υπάρχουν στην αγορά τα πλονεκτήματα της ενεργειακής εξοικονόμησης που θα μπορούσαν να προκύψουν από την βελτίωση των κτηρίων και βελτίωση όσον αφορά τα κόστη και την κατανάλωση. Να θυμίσω και τα όσα είπε χτες και ο αντιπρόεδρος Εύκοβιτς που υπογράμμισε ότι ε, είναι ανάγκη στο εγγύς μέλλον όχι μόνο να κατασκευάζονται κτίρια τα οποία να είναι αποδοτικά από άποψη ενέργεια, αλλά και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να ε, σχεδιάζουμε ευφυή e κτίρια και σπίτια που θα μπορούν να παράγουν ενέργεια, να αποθηκεύουν την, ε, ε, το περίσεμα, ας πούμε, για να μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθεί έρευνα και ανάπτυξη, να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και την έρευνα. Όσον αφορά και τελειώνω την χρηματοδότηση και τις, ε, τα κίνητρα στον τομέα αυτό, γιατί χρειάζονται ολοκληρωμένες προσπάθειες από όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία και είναι πολύ σημαντικό αυτά να είναι προσβάσιμα όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν την μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών της Ευρώπης. Τέλος, ένα σημείωμα όσον αφορά την βιομάζα που αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή μια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται πολύ στον τομέα της θέρμανσης, ε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η χρήση της επιφέρει και κάποιες αντιδείξεις. Κάποια, στη, κάποια είδη βιομάσας, ας πούμε, βιομάζες, ε, σημαίνουν σημαντική αύξηση των αερίων θερμοκηπίου και άλλα μικρά σωματίδια ε, που είναι ρήπη. Επίσης, ε, χρησιμοποιείται για διαφορετικούς όρου, σκοπούς. Για να συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο είναι σημαντικό να στοχεύσουμε μόνο στην βιώσιμη βιομάζα από άποψη περιβαλλοντική βιώσιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Ντάνκαν απουσιάζει, όπω και ο κύριο Σελίμοβιτ, η κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια τον εισηγητή συγγνώμη, για ε, μια σειρά από πολύ καλά σχόλια. Μιλάμε για το 50% της, των ενεργειακών αναγκών και ένα από τους πιο σημαντικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η ενεργειακή, απόδοση θα συνεισφέρει στην ε, οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μας βοηθήσει ταυτόχρονα και στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια μέσω της βελτίωσης αποδοτικότητας. Το πρόβλημα δεν είναι η στόχη όμως, όσο η εφαρμογή από πλευράς των μελών. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ότι διαθέτουμε πολύ λίγα χρηματοδοτικά μέσα για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων με ψηλή ενεργειακή απόδοση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ανακαινιστεί περίπου το 3% το όλων των κτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προσαρμοστεί. Ε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει ένα χρηματοδοτικό σύστημα μοντέλο ε, για την ανακαίνιση και των δημοσίων, κρατικών αλλά και των ιδιωτικών κτηρίων. Σε ό,τι διαφορά τη βιομάζα, η Κομισιόν λέει ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα μας έχει υποβάλει μέτρα, προτάσεις μάλλον, για την βιωσιμότητα της ε, χρήσης ε, βιομάζας. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία της Κομισιόν. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη βιομάζα προφανώς, αλλά ξέρουμε τι έχει φέρει ως τώρα η προώθηση των ε, βιοκαυσίμων τι συνέπειες είχε στο περιβάλλον. Οπότε λίγη προσοχή. Επιπλέον, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής παράδοξο στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Ο συνδυασμός ε, της παραγωγής ε, θέρμανσης και ψήξης θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όμως αυτό θα χρησιμεύσει σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς. Δεν υπογραμμίζεται πολύ συχνά το γεγονός όμως ότι υπάρχει έλλειψη χρηματοδοτικών μηχανισμών και ταυτόχρονα το γεγονός ότι έχουμε ε, σταθμούς παραγωγής ε, θερμικής ενέργειας με σημαντική αποδοτικότητα όπως καύση αποβλήτων κλπ. Αλλά δεν έχουμε ε, επαρκείς κανόνες για, τα, για τους σταθμούς ε, καύσης. η ποιότητα του αέρα, η κλιματική αλλαγή, η καύση των αποβλήτων, όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στις προτάσεις της Κομισιόν. Γιατί σχετίζονται μεταξύ τους και αυτό είναι και, θα είναι και το βασικό μας καθήκον τα επόμενα χρόνια ως Επιτροπή ΕΜΒΗ, ως Η νομοθέτηση απλώς δεν θα μας οδηγήσει στην επιτυχία των στόχων, χρειάζεται και σωστή εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άουκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Φιέλνερ για ε, το σχέδιο της νομοδότησής του. Είναι πάρα πολύ σαφές και στα περισσότερα σημεία συμφωνούμε ανεπιφύλακτα. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ξεκάθαρα γιατί εμβέλεια ε, προβλήματος ε, συζητάμε σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας έτσι όλα αυτά να λειτουργούν ε, τέλεια. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η ουδετερότητα ως προς την τεχνολογία. Τι εννοώ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παρενέργειες των εισαγωγικών αν γίνεται λόγος για τη Δανία, πολύ συχνά ακούμε και για τη Σουηδία ότι ε, έχουμε πολλά σπίτια με σόμπες. Εντάξει. Μπορεί και να χρησιμοποιείται ξύλο που είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αλλά ε, ε, αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, γιατί απελευθερώνονται αερούμενα σωματίδια και τα λοιπά στη Γανία. εμείς λατρεύουμε αυτές τις σόμπες, αλλά ξέρουμε και τη ζημιά κάνουν στην υγεία. Δεν είναι λοιπόν τα πάντα ρόδινα. Το ίδιο ισχύει και για τη βιομάζα. Και καλά κάνεις, Κρίστοφερ, και τα λες στη γνωμοδότησή σου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια πάρα πολύ καλή ε, μελέτη για την ε, αηφορία και τη βιωσιμότητα της ε, χρήσης της βιομάζας. τι γίνεται με τη χρήση των γεών, τι γίνεται με τα δάση, τι επιφάνειες θα χρειαστούν. Αυτά όλα θέλουν μελέτη. Και την πληρώνουν και τα τρόφιμα μετά. Δηλαδή καλλιεργούμε ε, φυτά ε, τα οποία είναι βρόσιμα για να καταλήγουν ε, στο ρεζερβόρ των αυτοκινήτων, το βιοκαύσιμο. Ωραία όλα αυτά για τη βιομάζα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι ζητήματα που χρειάζονται σωστή μελέτη, σωστή στρατηγική για να τα κάνουμε σωστά. Καλή η προθυμία και η συζήτηση με υψηλέ προδιαγραφές, υψηλέ απαιτήσει ε, και στοχοθεσία. Αυτό ισχύει και για την ε, βιομηχανία και είναι και υγιές αυτό γιατί μπορεί να επαφίεται σε αυτά που ζητούμε, να βασίζεται και να είναι μακροπρόθεσμη η προσπάθεια. Υπάρχουν και προοδευτικοί κλάδοι στην οικονομία που συχνά εκτοπίζονται από τις παλιές παραδοσιακές και παλιωμοδίτικες. Το είδαμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενδεχομένω να το δούμε και σε αυτόν τον κλάδο. Για την κυκλική οικονομία και την αξιοποίηση των αποβλήτων, νομίζω ότι στην Δανία είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στην αποτέφρωση των ε, αποβλήτων. Πυρομανείς είμαστε πρωταθλητές στο να καίμε σκουπίδια. Έχουμε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις που δεν εκπέμπουν σχεδόν καθόλου διοξίνη, αλλά ε, έτσι και με και πόρους, γιατί τα σκουπίδια είναι ε, πόροι. Η αποτέφρωση των αποβλήτων ε, δεν είναι πάντα η σωστότερη λύση για την ανακύκλωση και μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση και ψήξη από διάφορους κλάδους της οικονομίας και της βιομηχανίας. Και σε μια κυκλική οικονομία δεν μπορούμε να περάσουμε από τα και με τα σκουπίδια. Είναι πόρος το απόβλητο και εμεί πάμε και τα καίμε και τα χάνουμε. Και στην ε, ιεραρχία των αποβλήτων ε, ή την κυκλική οικονομία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό. Ελπίζω να συμφωνήσουμε σε όλα αυτά. Κρίστοφερ, ευχαριστώ πάντως για την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αφρόντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια στοιχεία για να συμπληρώσουμε την έκθεση του εισηγητή που νομίζουμε πως είναι πολύ καλή, αλλά ότι μπορεί να ενισχυθεί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι επενδύσεις που γίνονται για να μειωθεί η χρήση της, να αλλάξει η χρήση της ενέργειας σε βιομηχανικό επίπεδο είναι εκείνοι που δίνουν τους πιο σύντομους χρόνους ε, ανάμεσα στην επένδυση και την εφαρμογή και επίσης την, τους πιο γρήγορου χρόνους ε, ανάμεσα στην επένδυση και την μείωση της ζήτησης. Ε, επίσης θα πρέπει να θυμίσουμε μέσα από την έκθεση ότι θα πρέπει να είναι δεσμευτική η στόχη για την ενεργειακή επάρκεια σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης ε, καθώς επίσης και μια ενιαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ε, ε, ενεργειακών εξοικονομήσεων και της απόδοσης. δεν υπάρχει κάποιος κοινός τρόπος για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Έπειτα, για την ε, παραγωγή της θερμικής ενέργειας δεν συμφωνώ πολύ με τους συναδέλφους που μίλησαν πριν, γιατί για μας η καύση, ακόμα και με την ε, ανάκτηση της ενέργειας και ακόμα και με τη θέρμανση, δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη ε, μέσω και μακροπρόθεσμα, ούτε για τη διαχείριση των αποβλήτων, ούτε για την πρόθεση των εναλλακτικών ενεργειακών πηγών για την θέρμανση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κινούμαστε σε παράλληλες γραμμές. Μιλάμε για κυκλική οικονομία μία δηλαδή και μηδενικά απόβλητα, ένα σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν δηλαδή πλέον ε, τα απόβλητα και από την άλλη πλευρά μιλάμε για συστήματα παραγωγής ενέργειας που να μας επιτρέπουν και τη διαχείριση των αποβλητών. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά το όνομα το άλλο. Το η υπόθεση της βιομάζας ε, αναφέρθηκε από διάφορους συναδέλφους ε, και συμφωνώ με την συνάδελφο Άουκεν ότι η Κομισιόν πρέπει να μας δώσει κριτήρια βιωσιμότητας που αυτή τη στιγμή λείπουν. Δηλαδή θα πρέπει ε, να ε, αυτή η βιωσιμότητα να είναι σχετική για το σύνολο του κύκλου ζωής, όχι μόνο ε, τη στιγμή της κατανάλωσης αυτής της βιομάζας και επιπλέον, και εδώ συμφωνώ με τη συνάδελφο Άουκεν, όταν λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ε, συστήματα μείωσης των ρήπων όπως ε, τα σωματίδια και η σκόνη και να μην γίνεται μια γενικόλογη αναφορά στην ποιότητα του αέρα, πράγμα το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την αύξηση της χρήσης της βιομάζας για την θέρμανση των πόλεων. Θέλουμε επίσης να ε, υπογραμμίσουμε το θέμα της ε, θέρμανσης και της ψήξης. το συνδυασμό και το μεγάλο δυναμικό της γεωθ θερμικής δυνατότητας ε, που κατά κάποιο τρόπο ε, εξομαλύνεται έτσι η προσφορά της θερμικής ενέργειας, της, ε, ε τέλος, στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, αναφέρεται το και το θέμα της συνειδητοποίησης, της γνώσης, της ενημέρωσης των καταναλωτών που σήμερα ας πούμε ορίζουν ε, συχνά για μεγάλες ε, χρονικές περιόδους την θερμοκρασία με θερμοστάτες και χρησιμοποιούν μεθόδους που δεν είναι πάντοτε οι καταλληλότερες σε σχέση με την πραγματική απέτηση. Θα μπορούσε ας πούμε να να, να, να θυμίσουμε τον και να στηρίξουμε τις παλιές παραδοσιακές μεθόδους ψήξης ή θέρμανσης, να θυμίσουμε ας πούμε τον ανεμιστήρα τον καλό παλιό ανεμιστήρα που μπορεί να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του χωρίς να ρηπαίνει όπως ένα air condition. Κυρία Γκροστέτ, ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συνδέεται απόλυτα με τις συζητήσεις που είχαμε και χτες το απόγευμα με τον Αντιπρόεδρο Σεφκοβιτς. Πολύ συχνά υπάρχει μεγάλη απώλεια ενέργειας σε μη μονομένα κτίρια, κτίρια και πρέπει να Ε, το συζητήσουμε και να το αναφέρουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Αυτό τα δίκτυα είναι μια λύση που επιτρέπει σε αστικό πλαίσιο να χρησιμοποιηθεί η, θερμότητα που προκύπτει από την βιομηχανική παραγωγή ενός εργοστασίου. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα ε, Υπάρχει το θερμό, το, το ζεστό νερό που μπορεί να μεταφερθεί και λειτουργεί χωρίς καύσιμο. Ε, όσον αφορά την ασφάλεια ε, ανεφοδιασμού, τέλους είδους ε, ε, θερμάστρες λειτουργούν με βάση διαφόρων ειδών ενέργεια. Είναι αρκετά ευέλικτο σύστημα γιατί καλεί και χρησιμοποιεί διάφορες δυνατότητες. Ε, με πολλούς συναδέλφους μίλησαν για τη βιομάζα, την στερεή με το ξύλο, ναι, αλλά και υπάρχει εκπομπή σωματιδίων, άρα θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά αποδοτικές εγκαταστάσεις για να συλλέγουν αυτά τα σωματίδια, αλλά κανείς δεν αναφέρει το βιοαέριο. Το βιοαέριο επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω της μεθανοποίησης. Είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται από διάφορες φάρμες ε, αγροκτήματα στην Ευρώπη. Είναι μια πηγή. Και εδώ πρέπει να κάνουμε έκκληση στην κυκλική ε, οικονομία και είναι καλό να ενσωματωθεί και αυτή η δυνατότητα. Στην Ευχαριστώ. Λαχάη. Κύριε Αντελέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, δεν θα επαναλαμβάνω ε, και εγώ, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ. Ε, με κάλυψε. Θέλω να πω κάτι για τη ε, βιομάζα, το βιολογικό αέριο. Όπως είπε μόλις η κυρία Γκροστέτ, ε, είναι σημαντικό τμήμα και τομέα δραστηριοτήτων για τα αγροκτήματα και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη. Θα ήθελα όμως να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τι βάζουμε σε αυτές τις εγκαταστάσεις μεθανοποίησης, δηλαδή να μην είναι ό,τι να είναι ε, από απόβλητα ε, για να δημιουργήσουμε αυτό το βιολογικό αέριο. Έτσι, στη σύνθεση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική η χρήση και η ιεράρχηση των αποβλήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσουμε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. No Δεν έχει γνώμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρουσία. Good uh, uh, Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για τα σχόλια. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι σε σύγκρουση με τις προτάσεις μας. Συμφωνούμε με τα σχόλια των βουλευτών. Διαβάσαμε πολύ προσεκτικά και το προσχέδιο γνωμοδότης Επιτροπής. Να σχολιάσω απλώς εν συντομία τα βασικά σημεία των παρεμβάσεων. Πρώτον, αναγνωρίζουμε ότι η ψήξη και η θέρμανση είναι ε, ένας τομέας ε, πολύπλοκος, ε, δεν υπάρχει μία λύση για όλα. στην ανακοίνωσή μας εντοπίζουμε τις βασικές πτυχές με συγκεκριμένες δράσεις για κάθε μία οι οποίες όμως ε, θα εξαρτώνται από την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια του κλπ. Συμφωνούμε επίσης ότι χρειάζεται τα κτίρια μας να είναι πολύ πιο ενεργειακά αποδοτικά, να σταματήσουμε δηλαδή την ε, σπατάλη της ενέργειας, η ανακαίνιση των κτηρίων είναι πάρα πολύ σημαντική και σίγουρα θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και κρατικά και ιδιωτικά κονδύλια. Γι' αυτό θα πρέπει και οι κρατικοί φορείς και οι ιδιωτικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην, στο μεγάλο αυτό έργο της ανακαίνησης, ενεργειακής ανακαίνησης των κτηρίων. Και ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ευφύ τρόπους χρηματοδότησης. Ανακαίνιση λοιπόν και νέες τεχνολογίες στην κατασκευή των κτίριων είναι απαραίτητες και σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε πρώτη προτεραιότητα στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτίριων. Όλα αυτά συνδέονται προφανώς με το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών και η ενεργειακή αποδοτικότητα προφανώς είναι ένας από τους ε, πιο κατάλληλους τρόπους ε, να χαλιναγωγήσουμε το ενεργειακό κόστος. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με τα απόβλητα και την κάψη τους. Και εδώ προτείνουμε πιο δραστικές πολιτικές μέσω την, ε, της χρήσης της ενέργειας ε, θέρμανσης και ψήξης που προέρχεται από βιομηχανική παραγωγή. Ε, αυτό δεν αποτελεί κάψη των αποβλήτων. Η κάψη των απολύτων αποβλήτων θα παραμείνει ως ξεχωριστή μέθοδος. Αυτό που λέμε είναι ότι υφίσταται δυνατότητα ανακύκλωσης αποβλήτων βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, ακόμα και από τη γεωργία ενδεχομένω. Υπάρχει αυτό το δυναμικό, δεν ξέρουμε ποιο είναι, πόσο είναι, είναι μεγάλο. Αυτό που επιθυμούμε είναι να ερευνηθεί και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το δυναμικό θα ήταν καλό για την βιομηχανία, ε, για τη μείωση του κόστους και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν θα έσπροχνε την, ε, δεν θα οθούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγει περισσότερα απόβλητα. Η βιομηχανία πάντοτε θα έχει κάποια ανάγκη χρήσης ε, ενέργειας από άνθρακα, τουλάχιστον για πολλά χρόνια ακόμα. Το ίδιο και στη γεωργία. Θα πρέπει να δούμε ποιο πόσο μπορούμε να ανακυκλώσουμε και αν υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό, γιατί να το χάνουμε, γιατί να το σπαταλάμε. Χρειάζεται όμως έρευνα. Σε ό,τι αφορά την βιοβιωσιμότητα, Η Κομισιόν σκοπεύει, όπως είπαμε, να υποβάλει προτάσεις για κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα. Η, ιδιαίτερα η βιομάζα, επίσης ε, η χρήση βιομάζας ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές μπορεί να αποτελέσει και κίνδυνο για την υγεία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε τα σχόλιά σας. Η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν επίσης ε, ε, θέτει ως στόχο την βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της ενημέρωσης του. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από τους κατασκευαστές, τους εργολάβους, τους ιδιοκτήτες, μετά τους ενοικιαστές και προφανώς τις κρατικές αρχές. Θα πρέπει όλοι αυτοί να είναι ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες και τα ωφέλη στην υγεία και αλλού που μπορεί να προκύψουν με τη χρήση τους. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, θέρμανση ε, εξ και την ψήξη εξ είναι ένα τομέα στον οποίο έχουμε εντοπίσει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πιο σοβαρά. Ενδεχομένως στην οδηγία, στην αθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποιες διατάξεις γι' αυτό. Η χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών στην εξαποστάσιο θέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομίες ενέργειας και στην πρόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακριβώς διότι ορισμένες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι οικονομικά ε, αποδοτικές ε, αν χρησιμοποιηθούν μόνο σε ε, συγκεκριμένα λίγα κτίρια, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εξαποστάσεως θέρμανση που παρέχει θέρμανση ε, από ένα κεντρικό σημείο για μια ολόκληρη περιοχή. Όχι λοιπόν σε μεμονωμένα κτίρια. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τα σχόλια σας, τα λάβουμε υπόψη. Πρόεδρος, ο λόγος στον εισηγητή. Παρακαλώ συντομία. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς με χαρά ακούω ε, τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει για συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση ολόκληρων περιοχών με ε, θέρμανση θέρμανση με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων κτλ. Υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος αυτής της ε, δυνατότητας, δεν αξιοποιείται απολύτως. Πολλά τα καλά σχόλια. Διαπιστώνω ότι θα χρειαστεί να συζητήσουμε για τη βιομάζα αυτό δεν είναι κάτι το νέο, είναι περίπλοκη η κατάσταση όμως. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα όπου δημόσια κονδύλια και ε, καμπάνιες ε, που αγωνίζονται να παραμείνει το τοπίο ανοιχτό και ε, να μην μας κατακλείσουν τα δάση που ε, κινδυνεύουν να κυριεύσουν όλη τη χώρα. Ξέρω ότι σε άλλες χώρες διαφέρει η κατάσταση. Η βιομάζα είναι τα δύο τρίτα των ανανεώσιμων που χρησιμοποιούμε σήμερα. Είναι τεράστιο το ποσοστό στο μείγμα. Και η αύξηση της βιομάζας θα είναι κρίσιμη στο μείγμα αυτό το ενεργειακό των ΑΠΕ. Αλλά και για τα απόβλητα και για τη βιομάζα θα ήθελα να σκεφτείτε μέχρι να κάνετε τις απολογίες το εξή. Δεν μπορούμε να, να μπούμε σε αυτή την ε, ε, συζήτηση έχοντας απέναντι, έχοντας αντίπαλο το βιολογικό αέριο τη βιομάζα γιατί έτσι θα κερδίσουν τα ορυκτά καύσιμα. Τα ανανεώσιμα ή ανανεώσιμε πηγέ έχουν προβλήματα και η βιομάζα και τα απόβλητα, αλλά μην ξεχνάτε τι σημαίνει ο άνθρακα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και δε συμμαζεύεται. Εκεί είναι τα πραγματικά προβλήματα και τα μεγαλύτερα. Δεν είναι αντίπαλοι μα ε, οι ανανεώσιμε ή κάποιο είδο ανανεώσιμη ε, πηγή ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε αυτό το κλάδο της χρήσης ξυλίας για ε, θέρμανση αποβλήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να θυμίσω τώρα το χρονοδιάγραμμα προθεσμία κατάσταση απολογιών. Μόνο στα αγγλικά οι τροπολογίες. 26 Μαΐου. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 21 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί. Στην Επιτροπή Ήτρε 12 Ιουλίου και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβρη. Μπορεί να τελειώσει εδώ αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο που λέει ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα. ο διαπλαίσιο για τα απόβλητα και τα απορρίμματα συσκευασίας. έχουμε συμφωνήσει να έχουμε μόνιμη ανταλλαγή ε, απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Σήμερα είναι η πρώτη φορά ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή της παρεμβαλλοντικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία πλαίσια, όπως είπαμε, για τα απόβλητα και τα απορρίμματα συσκευασία. Οι συνάδελφοί μας έχουν υποβάλει 23 ερωτήσεις που επικεντρώνονται σε διάφορα προβλήματα εφαρμογής και μέτρα, διαλογή των αποβλήτων, των απορριμμάτων, ε, υποπροϊόντα, κριτήρια μη παραγωγής και πρόληψης ε, απορριμμάτων, ε, διάφορα ειδικά θέματα αύξησης, συνειδητοποίησης κτλ. Τώρα, προτείνω να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει ε, σε κάθε ομάδα ε, ερωτήσεων γύρω στα 10 λεπτά για την πρώτη και τη δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους συντάκτες των ερωτήσεων για να κάνουν επερωτήσεις, αν θέλουν. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα και τις προκλήσεις της εφαρμογής για τις ερωτήσεις 1 έως και 6. Να μας απαντήσετε μαζί όλα αυτά τα ερωτήματα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία των ερωτήσεων και απαντήσεων. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρευρίσκεται ο κύριος Τζομπάρ Ντορντέα και ο κύριος Αντάουσκας. Έχετε το λόγο. Uh, uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση θα κάνω κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις και μετά θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο της Τούτης. Κάποιες παρατηρήσεις για να τοποθετήσουμε στο πλαίσιο τις προσπάθειες εφαρμογής ε, το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων ε, από πλευράς Κομισιόν και TGA περιβάλλον. Ξέρετε, η Κομισιόν έχει μοναδικό και ουσιαστικό ρόλο στην επίβλεψη της εφαρμογής ε, και της εκτέλεσης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι απόσπαστο τμήμα της εθνικής νομοθεσίας και τα κράτη-μέλη και οι δημόσιες αρχές τους καλούνται να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει την ε, δυνατότητα να επιβλέψει την εφαρμογή από πλευρά των κρατών μέλων και θα έλεγα <clears throat> ότι από στρατηγικής ε, άποψης η Κομισιόν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εφαρμογής ε, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της εφαρμογή τη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων επί τριών βάσεων. Πρόθεση της συμμόρφωσης, τριών αξώνων μάλλον. Η σωστή λειτουργία και η συνεργασία με τα κάτι μέλη για την εφαρμογή, η παροχή οικονομικής στήριξης για τη συμμόρφωση και τρίτος άξονας είναι η επιβολή των κανόνων όταν οι προσεγγίσεις συνεργασίας δεν λειτουργούν. Για την πρόθεση της συμμόρφωσης, η Κομισιόν, λόγω των πολλών ετών εργασίας επί της εφαρμογής και στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, έχουμε σαφή γνώμη για το ποια είναι τα αίτια της ε, Προβληματική εφαρμογή. Κάποιες φορές πρόκειται για έλλειψη πολιτική βούλησης, άλλες φορές έλλειψη οικονομικών πόρων, ενώ άλλες φορές πρόκειται για περίπλοκες ρυθμίσεις στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων. Όμω πιστεύουμε ότι με την ανάληψη του τωρινού συνόλου επιτρόπων, καθηκόντων, ανάληψη καθηκόντων του σημερινού συνόλου των επιτρόπων, πιστεύουμε ότι έχει δοθεί περισσότερη έμφαση στην εφαρμογή και την εκτέλεση και ότι και εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να ξεπεράσουμε τον τεχνικό διάλογο με τα κράτη-μέλη, που είναι απαραίτητο βέβαια, αλλά και να επιστήσουμε πολιτική προσοχή στι κυρίε προκλήσει εφαρμογή και στον τομέα τη διαχείριση αποβλήτων. Επίση, πρέπει καλύτερα να ενημερώσουμε το κοινό για αυτές τις προκλήσεις και να προσφέρουμε ευρύτερη εικόνα ώστε όλοι οι ε, υπουργοί και κοινή γνώμη η <coughs> πολιτικοί εδώ και στο Συμβούλιο να καταλάβουν τις προκλήσεις. Πολιτικό προφίλ λοιπόν της εφαρμογής με την υιοθέτηση μέχρι το τέλος του μήνα πριν τις 31 Μαΐου δηλαδή, μιας ανακοίνωσης όπου θα εξηγούμε το πλαίσιο για μια νέα πρωτοβουλία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή και λέγεται αναθεώρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πριν ε, το τέλος του μηνός και μάλιστα μέχρι το τέλο του έτου θα έχουμε και εκθέσεις ανά χώρα και για τι 28 χώρε που δεν θα ασχολούμαστε μόνο με τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και με τα μείζωνα θέματα περιβαλλοντική πολιτική. Και πώ τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται στι υποχρεώσει του και συμμορφούνται ε, στην κείμενη νομοθεσία. Η διαχείριση των αποβλήτων και η κυκλική οικονομία γενικότερα θα μας απασχολήσει και θα καλύψει ένα σημαντικό ε, πεδίο και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη ε, μας για το πάγιο ενδιαφέρον τη Επιτροπής σας ε, σε θέματα εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Το δεύτερο τώρα, πεδίο όπου συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη είναι χορήγηση κονδυλίων και υποστήριξη για τη διαχείριση των αποβλήτων, για να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει τα κράτη-μέλη. Πριν πούμε σε λεπτομέρειε ε, για την προηγούμενη πολιετή ε, προγραμματική περίοδο, ε, πρέπει να πω ευθύ εξ ότι τα κονδύλια που προσφέρονται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για αυτό το λόγο δεν είναι αρκετά σε ε, σύγκριση με τις ανάγκες των κρατών μελών. Αυτό είναι γεγονός και ισχύει και για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως και αλλού. Αλλά ε, το θέμα δεν είναι να χρηματοδοτηθεί η συμμόρφωση 100% ε, στα περιβαλλοντικά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα πρέπει και τα κρατημέλη και οι περιφέρειες να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να δεσμευθούν συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης της υποδομής για τη διαχείριση των αποβλήτων. Σήμερα λοιπόν θα έλεγα ότι η σωστή διαχείριση αποβλήτων είναι αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες κοινωνίες μας. Θα ήταν αδιανόητο να έχει κανείς ε, σωστές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων μόνο στις πρωτεύουσες. Παντού χρειάζεται αυτό σε όλα τα αστικά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι εκ των όνων και προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη μας. Έρχομαι τώρα ε, στην υποστήριξη που δώσαμε πέρα από την οικονομική την περασμένη περίοδο ε, προγραμματισμού 2007-2014 ήταν 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής για τις επενδύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων. Πολλά κράτη-μέλη που επωφελήθηκαν από τη χρηματοδότηση αυτή, έκλεισαν τις ε, χιτά που δεν ήταν σε σύγχρονες προδιαγραφές, έχουν αυξήσει τη διαλογή ε, για βίο αποσπόμενα και ανακυκλούμενα ε, απόβλητα και έχουν φτιάξει τις εγκαταστάσεις έκλεισαν χωματερές δηλαδή. Και έχουν διαχειριστεί εκεί τα κονδύλια. Σε ορισμένα από τα πιο καινούργια κράτη-μέλη πάνω από 10% ήταν ε, στη Βουλγαρία, Σλοβενία και Πολωνία αυτά. Ε, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020 η χρηματοδότηση είναι λίγο χαμηλότερη, όχι πάρα πολύ όμως, μην νομίζετε, είναι 5,5 δις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τα απόβλητα. Δύο είναι οι μοχλοί που χρησιμοποιούμε για την πίεση. Τα κράτη-μέλη για να χρηματοδοτηθούν ε, θα πρέπει να πληρούν κάποιους όρους. Υπάρχει μια ε, εξάντε αιρεσιμότητα, το γράφουν αυτά οι κανονισμοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα χρησιμοποιεί ως μοχλούς, αλλά και εξακολουθεί να πιέζει τα κράτη-μέλη για να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Εδώ θα θυμίζα ότι η ε, εξάντε αιρεσιμότητα, τα προπετούμενα δηλαδή, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλη του έτους. Το 2017 θα είναι μια χρονιά ευαίσθητη και λεπτή γιατί θα έρθει να αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια κράτη-μέλη ανταποκρίνονται σε ποια προαπαιτούμενα. Ο δεύτερο μοχλό στο μέσο πίεση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι τα έργα που προτείνουν τα κράτη-μέλη για νέα χρηματοδότηση θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Άρα δίνουμε προτεραιότητα σε ε, δραστηριότητες στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το δει αυτό με τρόπο πάρα πολύ αυστηρό για να χρηματοδοτεί νέα, ε, νέες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των υπολοιπόμενων αποβλήτων. Συνάδελφος θα σας τα πει περισσότερα αυτά, σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι από τα διορθωτικά ταμεία για τα απόβλητα. Στην τρέχουσα περίοδο τα περισσότερα κονδύλια θα πάνε στην Πολωνία, Κροατία, Σλοβακία και Ουγγαρία. Of the ε, ε, Στο παρόν στάδιο του προγραμματισμού δεν έχουμε την πλήρη ενημέρωση αν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν όπως έχει σχεδιαστεί τα κονδύλια αυτά στα προγράμματα. Ε, από την 1η Ιουνίου θα έχουμε αυτή την πληροφόρηση και θα αρχίσουμε να την αξιολογούμε. Και μέχρι τα τέλη του έτους θα πρέπει κανονικά να είμαστε σε θέση να ε, σας ενημερώσουμε περισσότερο. Στην Επιτροπή και τα αξιότιμα μέλη της αν ε, θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ένα τρίτο σκέλος και θα σταματήσω με αυτό είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, επιβολή των κανόνων. Σύντομα, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος διαχειρίζεται το 20% ε, των προσφυγών επί παραλήψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σοβαρό αυτό αρκετά, το 1 πέμπτον. Το 1 πέμπτον ε, έχει να κάνει με την επιβολή ε, των κανόνων που ισχύουν για τη διαχείριση των αποβλήτων. Καταλαβαίνετε με δύο λόγια πόσο σημαντικό είναι και πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε στη συμμόρφωση με ε, τη νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων. DG, ε, environment. Στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει γίνει και μια ερώτηση για το κατά πόσο οι ανθρώπινοι πόροι μας φτάνουν. Τώρα, τι να σας πω. Χαιρόμαστε που κάνετε αυτή την ερώτηση. Απάντηση έχει ως εξή. Στα πλαίσια της Ευρώπης των 28 κρατών μελών και με αυτά τα περίπλοκα θέματα που έχουμε στην νομοθεσία για τα περιβαλλοντικά, οι ανθρώπινοι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας είναι και σαν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τα ίδια συμβαίνουν. Ανεπαρκής δηλαδή. Πότε δεν θα έχουμε αρκετό κόσμο για να χειριστούμε αυτά τα θέματα, για να ε, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες και όλες τις προκλήσεις. Θα ήθελα όμως να σας επιστήσω την προσοχή στο έξη: Η εφαρμογή και η επιβολή ακόμα της νομοθεσίας δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως σας είπα και στην αρχή της τοποθέτησή μου, ε, είναι μια υπευθυνότητα αυτή με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, η παρακολούθηση, η εποπτεία ε, στο βαθμό που μας αναλογεί γίνεται με σωστό τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ε, ουσιαστικός αντίκτυπος επί τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε αυτή τη μικρή ακρόση. Να συνεχίσω τα λόγια του συναδέλφου μου. Πολλές φορές ε, υπάρχει η παρερμηνία ότι η τα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα είναι υπερβολικά περίπλοκα. Ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να τα μεταγράφουν. Είναι δική του ευθύνη, γιατί κυρίω πρόκειται για οδηγίε. Ε, η οδηγία για τα πλαίσιο για τα απόβλητα από την άλλη μεριά είναι η πιο απλή ενδεχομένω, που περιλαμβάνει γενικέ αρχέ. Και ποτέ η ερμηνεία της οδηγίας αυτής δεν αποτέλεσε εμπόδιο. Οπότε ε, η εφαρμογή είναι μεν προβληματική εξαιτία πολλέ φορέ έλλειψη πολιτική αποφασιστικότητα και οράματο. Δεύτερον, ε, εξαιτία του ότι νέε υποδομέ θα πρέπει να προγραμματιστούν πολύ νωρίτερα. Τρίτον, ε, ανάγκη να έχουμε χρηματοοικονομικά εργαλεία παρκή. Τέταρτον, Υπάρχουν αλλαγέ στη συμπεριφορά ε, ιδιωτικών και δημόσιων αρχών και οργανισμών και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και πέμπτον, ε, προβλήματα στην παρακολούθηση τη εφαρμογή και την επιβολή του νόμου. Ε, σε σχέση με τους στόχου του 2020 υπάρχουν λοιπόν αδυναμίες, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα 4-5 χρόνια να συμμορφωθούν και κάνουν βήματα. Οπότε είμαι αισιόδοξο. Πώ τι βοηθούμε, πώ βοηθούμε τα κράτη-μέλη από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίες επί παραβάση δεν λύνουν το πρόβλημα εύκολα. Ε, πρώτον διότι είναι καθυστερημένες και έχει ήδη γίνει ζημιά. Οπότε εστιαζόμαστε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη δίνοντα τους τεχνική συνδρομή να αλλάξουν τις πρακτικές τους. Ε, έχουμε πρωτοβουλίες πρόθεσης της συμμόρφωσης και βέβαια μέσω χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτουμε. Ε, προτιμούμε να χρησιμοποιούμε την προεδρευτική του καρότου δηλαδή και όχι του μαστιγίου. Ε, έχουμε πολλά χρηματοδοτικά μέτρα. Ε, έχουμε διάφορα μέτρα είπαμε. Πρώτον την πρωτοβουλία προώθησης της συμμόρφωση. Βοηθάμε τα κράτη μέλη με τα προγράμματα διαχείρισης. Ε, πρόσφατα αξιολογήσαμε 18 το ε, τα συστήματα δημοτικής διαχείρισης προβλήματος σε 18 κράτη-μέλη. Δεύτερον, σε συνεργασία με την υπηρεσία περιβάλλοντος, αξιολογούμε το πώς έχει εφαρμοστεί το κάθε κοινό σε κάθε κράτος μέλος και πώς έχει προχωρήσει σε σχέση με τις μόρφωσες στόχους. Η επόμενη έκθεση που θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη θα είναι έτοιμη στην αρχή του επόμενου έτους. Τρίτον, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω διαφόρων τρόπων, πλατφόρμες, εκδηλώσεις κλπ. Τέταρτον, εξετάζουμε τη συμμόρφωση της νομοθεσίας επισήμως και πέμπτον, μέσω νομικών διαδικασιών. Προσπαθούμε πάντοτε να βοηθούμε τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συλλογή και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Ε, και ε, η, επίσης ε, προβλέπουμε πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα για να στηρίξουμε, όπως για παράδειγμα το Horizon 2020, ε, το, την ε, στατικές επενδύσεις, την εταιρική σχέση για τις στατικές επενδύσεις. Ε, έχουμε μέτρα υποστήριξης καινοτομίας, ε, για, για το μοντέλο κυκλικής οικονομίας κλπ. Και προτείνουμε και ένα πειραματικό πρόγραμμα για να εντοπιστούν ενδεχόμενες ε, κανονιστικές, ε, ενδεχόμενα κανονιστικά εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν. Χρειαζόμαστε αρκετά εργαλεία και με αυτά τα εργαλεία, με τι κατάλληλε πολιτικέ, τα κράτη-μέλη μπορούν να σημειώσουν πρόοδο πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, η Σλοβενία αύξησε το, την ανακύκλωση από το 40% στο 60% σε τρία χρόνια. Σε μόνο τρία χρόνια. Ε, χρειάζονται όμω χρηματοοικονομικά μέσα και εμπειρία από τα πιο εμπειρά κράτη-μέλη. Και η εμπειρία αυτών των κρατών δείχνει ότι αυτά τα εργαλεία, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, είναι απολύτω σημαντικά για να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανακύκλωσης και της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα όργανα είναι, μέσα είναι ε, σταδιακά ε, τέλη καύσης και ε, ταφής, ε, ε, το να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες άμεσα υπεύθυνους για τα απορρίμματα τα οποία ε, δημιουργούν. Τρίτον, τέλη ε, ανακύκλωση και διαχωρισμού. Τέταρτον, επιβάρυνση αυτών που εμπορεύονται τα προϊόντα και θέλουν τα προϊόντα στην αγορά όταν αυτά τα προϊόντα δημιουργούν απορρίμματα στη χρήση τους. Η εμπειρία δείχνει ότι υψηλά τέλη ταφής είναι εργαλείο για να περάσουμε σε άλλους τρόπους διαχείρισης. Και επίσης πάνω από 70% των κρατών μελών ε, εφαρμόζουν συστήματα ε, ε, τελών που είναι αναλογικά με το όγκο των απορριμμάτων που παράγει ο κάθε καταναλωτής. Ε, θα κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση στο τέλος, μέχρι το τέλος του χρόνου. Στις προτάσεις για τα απορρίμματα όμως προτείναμε να καταργήσουμε την υποχρέωση έκθεση κάθε τρία χρόνια, διότι δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για να αξιολογήσουμε το που βρίσκεται κάθε κράτος μέλος. Οπότε προτείνουμε στα, στο μέλλον τα κράτη-μέλη να δίνουν στατιστικά στοιχεία μόνο για τους στόχους. Όμως, τα στατιστικά, αυτά τα στοιχεία δεν θα είναι η μόνη πηγή πληροφοριών για μας. Έχουμε πολλά εργαλεία, όπως είπα, στα ε, χέρια μας ε, για, την, για της εκθέσης μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I don't know if, uh... Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν να υποβάλουν Φλόρεντ, Φλόρεντς, Πιετικάινεν. είναι να... another time. Want to Θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Φλόρεντ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Παίρνω το λόγο γιατί είναι και το αγαπημένο μου θέμα, όπως γνωρίζετε. Έχω ένα πρόβλημα εδώ οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άνθρωποι συμπαθείς και έξυπνοι, αλλά όλα αυτά που μας είπατε σήμερα δεν μας ε, προχωράει ούτε σπίθαμη. Αυτά ακριβώς τα ίδια που είπατε θα μπορούσατε να τα είχατε πει και πριν από 10 χρόνια. Και ότι έχετε ακόμα πέντε χρόνια για να φτάσετε στους στόχους Μα το ξέρουμε εδώ και 10 χρόνια ότι μέσα σε μια πενταετία πρέπει να έχουμε φτάσει στους στόχους. Και αν διαβάσετε όλες τις μελέτες, τότε θα ε, δείτε πόσο θα σας πικράνουν όλα αυτά που θα διαβάσετε. Και δεν μιλάω για τις νέες χώρες και για τις παλιές και για τη δική μου τη χώρα την ίδια. Ε, δηλαδή, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό μας λέτε εδώ πέρα διάφορα πράγματα τα οποία δεν μας βοηθάνε καθόλου και δεν προχωρούν καθόλου την υπόθεση ούτε σπίθαμι ούτε ρούπι. Εγώ θα ξαναδιαβάσω αυτά που μας είπατε για να καταλάβω τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και των νόμων και δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το καθήκον. Το κατανοώ αυτό που λέτε ότι δεν έχετε προσωπικό ο Ποτότσινγκ φίλο που όποτε τον έβλεπα μου το έλεγε ξανά και ξανά. ενα να τα λέτε πιο δυνατά, να τα φωνάζετε αυτά περισσότερο, ότι δεν έχετε κόσμο. Και πού βρίσκεται το κουράγιο και το θάρρος. Τώρα να μας ε, προτείνετε την κυκλική οικονομία. Πολύ καλή έκθεση, δεν λέω, αλλά ξέρετε ότι τα θεμέλια στα οποία θα βασιστεί αυτό είναι σαφρά. 30-40% έχουν εφαρμοστεί άλλε οδηγίες. Καλά, κάποιο λίγο παραπάνω, κάποιο λίγο λιγότερο. Πραγματικά με εκπλήσει αυτό. Και ο Πίτροπός σα και όλοι οι άλλοι υπεύθυνοι θεωρούν ότι πω πω αυτό είναι τώρα super μπαλαντέρ, τζόκερ. Και αν κοιτάξετε πίσω από την κουρτίνα θα δείτε αμάν τι κάναμε. Πρέπει να κάνουμε πολύ λιγότερα και πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερα, πολύ πιο συγκεκριμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, το παρακολουθούμε. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Η πολιτική των υδάτων στο Ρήνο, ο οποίος ως γνωστόν ρέει από τη, Γαλλία προς τη Γερμανία αν πάτε στο ΚΕΛ, στα σύνορα με το Στρασβούργο και πάρει ένα δείγμα, θέλει να πάρει η Κομισιόν δείγμα από τη Γερμανία, πρέπει να στείλει ε, ε, επιστολή στο Βερολίνο αν επιτρέπετε. Το Βερολίνο θα σας πει να ρωτήσουμε τη Ρινανία Παλατινάτο που είναι το λόγο κρατήριο και θα σας απαντήσουμε. Μέχρι να σας απαντήσουν ναι, θα έχει περάσει και ένα εξάμεινο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν έτσι διαχειρίζεστε εταιρεία, θα βάλτε λουκέτο. Μην μας φαίνεται τόσες νέες εκθέσεις. Κοιτάξτε τις παλιές. Στη Γερμανία, κοιτάξτε τι γίνεται. Η οδηγία για τα νητρικά, για να μην μιλήσω για άλλη χώρα. Αλλά κάντε τα καθήκοντά, μάλλον τα κράτη... Στο σχολείο ε, αν δεν έκανα τα μαθήματά μου, θα είχα μείνει στην ίδια τάξη. Δεν θα έπαιρνα ποτέ προαγωγή. Με κυνηγούσε κάθε εβδομάδα ο πατέρα μου, βάζει φωτιά στην καρέκλα. Παλουκό σου να διαβάσει. Δηλαδή, ε, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Ik heb een optimistische commissie inderdaad. Άκουσα και εγώ μια αισιόδοξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η αισιοδοξία φυσικά είναι ηθικό καθήκον. Moral duty το λένε οι Άγγλοι αυτό. Αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Και συμφωνώ με τον κύριο Φλόρενς. Για να γίνει πραγματική πρόοδος, αυτό που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά τι φταίει που υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορές και ε, αποκλίσεις στην ε, εφαρμογή της ίδιας μας της νομοθεσίας, των οδηγιών μας. Και σε ό,τι αφορά αυτό, δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις σας επαρκώς. Έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια για να ε, καλύψουμε τους στόχους. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά είναι λίγο αισιόδοξη ως προς αυτό. Και έχω την εντύπωση ακόμα ότι πάρα πολύ ε, παραμένουμε στη λογική των αποβλήτων. Τι εννοώ. Ε, συζητάμε συχνά ε, ε, τα αποβλήτα και για τη λογική ε, που μας διέπει που είναι πώς θα ξεφορτωθούμε τα απόβλητα. Θα πρέπει να το δούμε αλλιώ. ως φυσικούς πόρους, ως προς την ανταγωνιστικότητά μας. Θα πρέπει να εξακολουθούμε να προβληματιζόμαστε αν μπορούμε να επιτρέπουμε τόσο πολύτιμη φυσική πόροι να χάνονται, γιατί και αυτό είναι τα απόβλητα. Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα. Άρα, στην πράξη θα πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ε, πού οφείλονται οι διαφορές και από πού ε, προέρχονται. Και έχω την εντύπωση ότι το θέμα είναι η πολιτική βούληση εδώ που λείπει. Αυτό που θέλουμε είναι να αναλάβουν την ευθύνη τους και να δείξουν προθυμία και τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία και τα νομοθετικά στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να δουλέψουν. Εγώ προέρχομαι από τη Φλάνδρα, κατάγομαι, όπου μπορώ να το πω, είναι από τους πρωτοπόρους και ε, ε, έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις ε, στη διαλογή, στον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται η αποκομιδή των απορρίτων. Χρειάστηκε και χρόνο και πολιτικό θάρρος, αλλά τα καταφέραμε. Και είμαστε ε, μπροστά, έχουμε κάνει δεκαετίες ολόκληρες βήματα. Δεν είναι υπόθεση αυτή βράχη πρόθεσμη. Και είμαστε πραγματικά περήφανοι, νομίζω μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε πετύχει. Άρα, θα πρέπει να δείξουμε και σε άλλα και περιφέρειες ότι δεν ξεκινάνε από το μηδέν, δεν είναι μηδενική βάση. Υπάρχει εμπειρία από άλλους. Ας πούμε η Σλοβενία που είναι καλό παράδειγμα όντως, μπορεί να κάνει ε, πράγματα, γιατί υπάρχει τεχνογνωσία, πραγματογνωμοσύνη σε άλλες περιφέρειες στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να τα εφεύρουν από την αρχή και έτσι μπορεί να γίνουν άλματα καλά τα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ε, αρκέσουν. Και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση για να φτάσουμε εκεί. Γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί. Και να φροντίσουμε οι πόροι μας, αυτό το απόθεμα, αυτός ο πλούτος στο κάτω-κάτω να παραμένει στην Ευρώπη και έτσι θα είμαστε και λιγότερο εξαρτημένοι από άλλους για την ενέργεια και θα αυξήσουμε και θα διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον, πρόκειται και για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία και για την ανταγωνιστικότητα. Είναι πλούτο το σκουπίδι. Ευχαριστώ, κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες και τις, ε, ε, τα όσα είπαν οι συνάδελφοι στις προηγούμενες παρεμβάσεις. Αυτό μου επιτρέπει να είμαι πιο σύντομη. Είναι προφανές ότι έχουμε ενώπιόν μας σε μια νέα νομοθετική πρόταση που σίγουρα θα επηρεάσει και τους νέους στόχους ανακύκλωσης καθώς και άλλους φιλόδοξους στόχους. Είναι σαφές ότι σήμερα με τις ισχύοντες κανόνες είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους. Γι' αυτό θα πρέπει κάτι να γίνει. Ε, Είμαι ωστόσο αισιόδοξη για το γεγονός ότι μπορούμε να δουλέψουμε, πρέπει να δουλέψουμε, κυρίως πάνω στην πολιτική βούληση, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν αρκεί το να κάνουμε διαδικασίε κατά παράβαση, πρέπει να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν αυτέ οι μεγάλε διαφορέ και αποκλήσει. Όμω θα πρέπει να υπάρχει μια σαφή αρχή ότι δηλαδή θέλουμε να κάνουμε κάτι σοβαρά. Δηλαδή να, να ενεργήσουμε για, πάνω στην πολιτική βούληση στα σοβαρά. Γι' αυτό και ο μηχανισμός που προβλέπεται σε αυτή την πρόταση, το Early Warning System, θα πρέπει από πλευρά της Κομισιόν να το χρησιμοποιήσει μέχρι τέλος, όπως χρησιμοποιείται και στα οικονομικά ζητήματα. Συμμερίζομαι λοιπόν την αισιοδοξία της Κομισιόν, όμως πρέπει να υπάρχει η βούληση να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα. Ευχαριστώ. Τόρμπανς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους εκπρόσωπους της Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να έχω κάποιες διευκρινήσεις για δύο σημεία. Καταρχάς είπατε ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα και ισχυρότερο προφίλ της. Θα ήθελα πολύ να καταλάβω τι είναι αυτό το νέο ισχυρότερο προφίλ. Να πειτά, μιλήσατε για εξαιρετική αυστηρότητα σε σχέση με την ιεραρχία των αποβλήτων. Καταλάβαμε ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο. Μιλάμε για αλλαγέ, τεχνολογικέ αλλαγέ. Εσεί είπατε ότι θα είστε πολύ αυστηροί. <clears throat> Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άλλες κατευθύνσεις. Περισσότερο από τις 10 εντολές για τις ε, πλάκες του Μωυσή. Εγώ δεν τα συμπαθώ πολύ όλα αυτά τα άκαμπτα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Στρέφομαι στη Κομισιόν για απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω πρώτα στις παρατηρήσεις του κυρίου Φλόρενς. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί ότι η κατάσταση δεν είναι ρόδινη, αλλά δεν είναι και μαύρη. Γιατί αν δούμε την πρόοδο και τη δυναμική των όσων έχουμε στην Eurostat, των στατιστικών στοιχείων που έχουμε στην Eurostat, βλέπουμε θετική δυναμική. Η Σλοβενία είναι ένα καλό παράδειγμα. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι εξωσημείωτο το πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να προοδεύσει αν ε, ακολουθήσει τις σωστές πολιτικές. Είναι αλήθεια ότι κάποια άλλα κράτη-μέλη ωστόσο έχουν μείνει πίσω και η ταχύτητα με την οποία ε, θα πρέπει να πετύχουν τους στόχους του 2020 δεν είναι αρκετά γρήγορη η θελημένη αμφισημία ήταν ότι τα κράτη-μέλη επιτρέπεται να ε, ανταποκριθούν και να πετύχουν τους στόχους σύμφωνα με τέσσερις μεθόδους και αυτό είναι ευκολότερο. Σύμφωνα με μία μέθοδο δεν θα το τηρούσαν, αλλά ο νόμος τους επιτρέπει τέσσερις μεθόδους. Και αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Να, να, να, το σταματήσουμε, να εστιάσουμε σε μια μεθόδο ώστε πραγματικά να μπορούμε να συγκρίνουμε και να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Επιπλέον και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι πολύ μεγάλο μέρος των αποβλήτων είτε καίγεται είτε θάβεται. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνεται πια. Τα απόβλητα που καίγονται να μην μετρώνται σαν ανακυκλούμενα. Αυτό έχουμε προτείνει στην αναθεώρηση. Γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα και αυτά θέλουμε να διορθώσουμε με τη βοήθειά σας. Νομίζω ότι εν γέννη είμαστε σε καλό σημείο σε σχέση με τους στόχους του 2020, αλλά θα πρέπει κάποια, κάποια κρατημέλη λίγα δεν θα τα καταφέρουν και γι' αυτό πρέπει να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει επί τόπου. Και μέσω της έκθεσης που θα εκπονήσουμε του χρόνου, και αυτό θα είναι και η έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτούς που πραγματικά κινδυνεύουν να μην πετύχουν τους στόχους και να τους συστήσουμε και δράσεις. Δεν είναι ρόδινη όπως είπε η κατάσταση, αλλά δεν είναι και μαύρη. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Δημεσμάκερ για το υπέρβαση των αποβλήτων και αυτό φυσικά χρειάζεται πολιτικό θάρρος αλλά και όραμα και αυτό λείπει συχνά σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό. Η Φλάνδρα είναι πολύ καλό παράδειγμα, μακάρι να ήταν η ολόκληρη Ευρώπη έτσι. Αλλά Έχετε δίκιο επίσης ότι δεν υπάρχει λόγος να πειραματιστούμε και να κάνουμε λέτσι λάθη ε, εφόσον κάποιες χώρες και κάποιες περιφέρειες τα έχουν ήδη κάνει. Μπορούν οι χώρες να μάθουν από τα λάθη των άλλων και να προχωρήσουν άμεσα σε αυτό που είναι σωστό. Και αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις μέσω των διευθυντικών ταμείων θα ακολουθήσουν τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό εννοούμε ότι θα είμαστε σκληροί και αυστηροί. Ε, απέναντι στα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν ότι με την βοήθειά σας μπορούμε να διαδώσουμε αυτές τις γνώσεις για τις καλύτερες πρακτικές και επίσης συνειδητοποιούμε ότι πολλές από τις δυσκολίες που υπάρχουν είναι σε διοικητικό επίπεδο, διαχειριστικό επίπεδο. Εκεί εντοπίζουμε πολλές φορές τις δυσκολίες ε, στις δημοτικές αρχές και νομίζω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας προκειμένου να διαδώσει τη γνώση και τις πληροφορίες. Το καλύτερο θα ήταν ε, μια ομάδα δημάρχων από τις χώρες που έχουν υστερήσει ε, να ε, επισκεφθούν πόλεις που έχουν διαχειριστεί, έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και να μάθουν εκεί δεν αρκεί απλώς να εντοπίζουμε τις βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να πιέσουμε και τους πολιτικούς να τις χρησιμοποιήσουν. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Και το πρόγραμμα δράσης για την κυκλική οικονομία είναι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε αυτό το θέμα με πιο ευρύ πνεύμα, διότι το πρόβλημα σίγουρα δεν είναι μόνο τα απορρίμματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now we... Ευχαριστώ πολύ. Μπορούν τώρα να αρχίσουν οι απαντήσεις ε, της δεύτερης ενότητας ε, των ερωτήσεων. Επάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση για τη διαλογή και την χωριστή αποκομιδή των αποβλήτων. Είναι οι ερωτήσεις 7 έως 12 και αργότερα θα συνεχίσουμε. Χαίρομαι που είναι μεταξύ των πρώτων ερωτήσεων διότι η διαλογή ε, στην συλλογή των απορριμμάτων είναι βασικό σημείο κλειδί για την ανακύκλωση, για τη σωστή ανακύκλωση ε, και την ποιοτική ανακύκλωση. Ως γενικό κανόνα ο γενικός κανόνας υπάρχει ε, σύνδεση ε, ανάμεσα στην υψηλή, στα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και την διαλογή στην πηγή. Στα κράτη-μέλη όπου γίνεται σε ευρύ επίπεδο διαλογή στην πηγή, γίνεται και μεγαλύτερη ανακύκλωση, περισσότερη ανακύκλωση. Η οδηγία πλαίσιο για τα απορρίμματα είναι σαφή. τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεχωρίζουν μέταλλο, πλαστικό, χαρτί ε, μέχρι το, τέλος του 2015. Ε, εκεί βέβαια που οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά είναι εφικτό για να γίνει ποιοτικά η ανακύκλωση αργότερα. Αυτός είναι ο όρος. Όμως ε, η ρήτρα ε, εφικτότητας θα πρέπει να ερμηνευθεί ε, περιοριστικά και μέσα στους στόχους της οδηγίας. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να ερμηνευτούν υπό το φω τη συνολική οδηγίας. Υψηλή προστασία δηλαδή περιβάλλοντο ανθρώπινης υγείας και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτή η αρχή τη εξαίρεση λοιπόν μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί και ε, να, ε, μόνο σε πολύ απομακρυσμένα νησιά ή σε πολύ αεροκατοικημένε περιοχέ και βέβαια αντχόξερα, αναπερίπτωση θα πρέπει να αξιολογείται με βάση κάθε περίπτωση χωριστά. Υπό το, φως αυτού η Κομισιόν προτείνει η ίδια αρχή να εφαρμόζεται ε, και στην ε, ξεχωριστή συλλογή, στο διαχωρισμό δηλαδή κατά τη συλλογή ε, δύο απορριμμάτων. Στην πρόταση για τα απορρίμματα λοιπόν θα προτείνουμε ε, και αυτό το μέτρο. Ε, αν δεν συλλέξουμε και τα δύο απορρίμματα θα είναι δύσκολο να συμμορφωθούμε τους νέους στόχους. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτή τη υποχρέωση, έχουμε να πούμε τα εξή. Ε, πέρσι άρχισε να ε, τέθησε ισχύ, παρόλα αυτά ε, το παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που υστερούν πιο πολύ περισσότερο στην διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε, ζητήσαμε μια, αναθέσαμε μια αξιολόγηση πολύ πρόσφατα για να αξιολογήσουμε το πώς εφαρμόζεται αυτή η υποχρέωση 28 κρατημέλη και η έκθεση αυτή έδειξε σημαντικές διαφορές στην διαλογή στην πηγή, στις ε, πρωτεύουσε και συνολικά στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και κάποια ακόμα και καινούρια κράτη-μέλη, τα οποία συσύλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, ε, που πρωτοπορούν, για παράδειγμα, η Λουμπλιάνα. Ε, η οδηγία απαιτεί διαλογή στην πηγή και είναι εφικτό αυτό όταν υπάρχει πολιτική αποφασιστικότητα. Ε, και μάλιστα δεν είναι και τόσο ακριβό. Αυτό έχει αποδειχθεί. Ε, εκεί που οι υποχρεώσεις αυτές δεν τυχάνουν πλήρους συμμόρφωσης, ο λόγος είναι οι, λόγοι είναι οι, λόγοι που γενικότερα ε, οθούν τα κάποια κρατημένα να στη διαχείριση των απορριμμάτων. Χρειάζονται υποδομές που πολλές φορές δεν υπάρχουν αλλά πολύ συχνά χρησιμοποιούνται πόροι ταμείου συνοχής ενώ κάποια άλλα κράτη-μέλη μέσω τελών με βάση την αρχή ορυπαίνων πληρένει. Πάντως είναι σαφές ότι οι προσπάθειες εφαρμογής αυτής της υποχρέωσης θα πρέπει να ενισχυθούν. Αργότερα, μέσα στο 2016, θα ξεκινήσουμε την συνολική συγκριτική ανάλυση και σε αυτή την ανάλυση θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει με την διαλογή στην πηγή. Και όταν έχουμε πλήρη εικόνα, οι προτεραιότητες πρόθεση μόρφωσης θα πρέπει να ενισχυθούν και αυτές. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε πώς και πότε τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση απαλλαγή από την υποχρέωση. Τους ζητήσαμε να μας αναφέρουν, έχουμε από τα κράτη-μέλη να αναφέρουν τους όρους και τις συνθήκες με τις οποίες θα το κάνουν. Θα το δούμε ε, όταν πάρουμε τις απαντήσεις οι επενδύσεις στα, των, των, του Ταμείου Συνοχής είναι ψηλέ σε αυτό το επίπεδο και αυτό είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι συνάδελφοι θέλουν να απαντήσουν. Κανείς, ο κύριος Δεμεσμάκερ. Een goede gescheiden ophaling Βεβαίω είναι προπόθεση για καλή ανακήρυξη, σωστή διαλογή. Πριν από λίγου μήνε και εγώ προσωπικά ε, οργάνωσα μια τέτοια επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο, σε μια ε, μονάδα ανακύκλωση στο Λιμβούργο, στη Φλάνδρα, όπου ε, φάνηκε ξεκάθαρα ε, πως από μια πρωτοπόρα επιχείρηση ε, μπορεί να λειτουργήσει. Ε, θα ήμουν ε, περίεργος να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ορισμό, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχουν κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη μάλλον υποχρεούνται να κάνουν αυτή τη διαλογή όπου είναι αυτό σκόπιμο και δυνατό από τεχνολογικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς. Αυτό είναι μια ε, απέτηση, ένα προαπαιτούμενο ε, που μπορούν όμως να χρησιμοποιήσουν ε, κράτη, μέλη και περιφέρειες ως δικαιολογία ή παραθυράκι για να μην το κάνουν. Έτσι όπως το ορίζετε, υπάρχει αυτό συμβαίνει, έχετε καμία τέτοια ένδειξη. Ένδειξη δεν έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία, έχουμε κάποιες υποψίες. Στις 28 πρωτεύουσες κάναμε μελέτες και έχουμε κάποια ιδέα για το τι συμβαίνει. Αλλά επειδή είναι καινούργια υποχρέωση αυτή και πρόσφατη, δεν ε, έχει ζητήσει κανείς ακόμα να κάνει χρήση αυτής της εξαίρεσης. Δεν μπορώ παρά να τονίσω και το λέμε και στα κράτη-μέλη ότι θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα το ερμηνεύουμε πολύ περιοριστικά. Και δεν μιλάμε για διαλογή σε πολύ απομακρυσμένες περιφέρειες που δεν χρειάζεται αυτό γιατί δεν είναι πάρα πολύ συχνή η συλλογή, η αποκομιδή των αποβλήτων. Αλλά επειδή είναι λίγες αυτές οι περιφέρειες σχετικά και είναι πολύ λίγα και τα απόβλητα που παράγονται σε σχέση με το σύνολο, αυτό είναι που εννοούμε και μπορούμε να δεχτούμε. Αλλά γενικά στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαλογή και το λέμε και στις επιχειρήσεις. Υπάρχει τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να αναμίξει απόβλητα και στη συνέχεια να τα ξεχωρίσει, ας πούμε πλαστικό και μέταλλο, να τα μαζεύει ε, από κοινού και μετά να το ε, χωρίζει. Αν βάλεις όμως ε, χαρτί με υγρά απόβλητα, καταστρέφεις και τα δύο και είναι πόρος αυτό. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε. Τα κράτη-μέλη ξέρουν πώς συλλέγονται χωριστά τα απόβλητα, αν όχι μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Τον Ιανουάριο κάναμε ε, μια διάσκεψη στις πρωτεύουσες, ε, προβλήθηκε και από την τηλεόραση ε, και εξακολουθώ να στέλνω στους συναδέλφους που το επιθυμούν βέλτιστες πρακτικές από κράτη που το κάνουν ήδη για να εμπνευστούν. Βλέπω ότι στο Κοινοβούλιο έχετε και τους κατάλληλους ε, ε, κάδους ε, και για την ανακύκλωση. Κύριος Φλόρενς, θέλω να πω κάτι για αυτά τα πολλά νομικά αόριστα πράγματα. Αυτά συνήθω δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πάρα πολύ συχνά από το Συμβούλιο ω διατυπώσει, διότι το Συμβούλιο, λόγω τη αρχή τη ομοφωνία, τουλάχιστον πολύ συχνά, δεν θέλει σαφεί κανόνε. δεν δέχεται. Θολώνει τα νερά. Εγώ πάντα τα λέω αυτά φιλελεύθερες παραγράφους ε, και τα βάζει ε, έτσι στη διατύπωση όπου ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν. Υπάρχουν χώρες που έχουν τεράστιο ταλέντο στην ερμηνεία και η δική μου μεταξύ αυτών. Προσοχή λοιπόν, φοβού τα κράτη-μέλη. Και έχουμε και εκεί για έναν σύντροφο ο οποίος ε, ανακατεύεται, που είναι η βιομηχανία. Και αυτή δεν θέλει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Γενικά θολώνουν τα νερά, θέλουν ε, μεγάλες και αόριστες και γενικές ε, ρυθμίσεις και όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία τόσο καλύτερα. Εμείς θα έπρεπε να είχαμε πιο στενούς ορισμούς, πιο περιοριστικούς, αλλά ούτε στο Συμβούλιο θα βρουν πλειοψηφία αυτά, ούτε εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο. Yeah. Then you just want to add the question on this. Oh, προσθέσω μια ερώτηση. Για αυτήν την ε, ιδιαιτερότητα ε, της οδηγίας, ε, πόσα έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την ειδική διάταξη του Qualifier για να ξεφύγουν από τις υποχρεώσεις τους και γιατί η Κομισιόν προτείνει να εφαρμοστεί το ίδιο για τη νέα υποχρέωση συλλογής των βιοαποβλήτων και να μην το διαγράψει τελείως. Αυτή η ειδική διάταξη δεν υπονομεύει την ουσιαστική εφαρμογή ε, της απέτηση για χωριστή ε, συλλογή. Τόρβαλτ, μια σύντομη ερώτηση σε σχέση με την χωριστή συλλογή και τα αποκομιδή και τα νέα υλικά που βλέπουμε στην, στην βιομηχανία συσκευασία ε, όπου έχουμε σύνθετα υλικά που είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα κατατάξει. Και θα ήθελα να γνωρίζω τι είδους προσέγγιση έχετε σε σχέση με αυτά τα υλικά, τα σύνθετα υλικά. Thank you. We have not additional question and we ask and we ask uh, the Commission to answer. Να ζητήσω από την Κομισιόν να απαντήσει. Μάλιστα. Μάλλον δεν μπορώ να ρωτήσω να απαντήσω στις ε, παρατηρήσεις του κ. Φλόρενς. Πρόκειται για παρατηρήσεις που απευθύνονται προς άλλο θεσμό. Εγώ μόνο μπορώ να επαναλάβω πως η δική μας ερμηνεία είναι περιοριστική, ότι η εξαίρεση είναι εξαίρεση και δεν μπορεί να γενικεύεται. Και έτσι απαντώ και στην κυρία Άοκεν ότι Πιστεύω πως είναι θέμα αναλογικότητας εδώ, γιατί σε μερικές περιπτώσεις κάπου στο βορρά, ας πούμε στη Φιλανδία ή στα νησιά, όπου δεν υπάρχει μάλλον ανάγκη για χωριστή αποκομιδή, όπου δεν μπορεί πραγματικά κανείς δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα, αυτό, εκεί μπορεί να υπάρξει εξαίρεση, αλλά μόνο με πολύ πολύ περιοριστική έννοια. Δεν έχουμε όμως τις πληροφορίες ακόμα για το πού εφαρμόζεται αυτή η εξαίρεση. Ε, βλέπουμε δηλαδή περισσότερο ε, και εστιάζουμε περισσότερο το τι κάνουν ε, τα κράτη-μέλη γιατί Θέλουμε να δούμε μήπως ε, χρησιμοποιούν εκεί όπου δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν. Εγώ δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, γιατί ε, δεν νομίζω πως είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αυτό που θα πρέπει να δούμε περισσότερο είναι το αν είναι αποτελεσματική αυτή η συλλογή. Μπορεί να βάλεις ε, τέσσερα σκάδου στο κέντρο μιας πόλης και να πει ότι είναι χωριστή εκεί η συλλογή των ε, αποβλήτων. Ε, θα πρέπει όμως να είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ώστε τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να εφαρμόζουν εξαιρέσεις όπου και νομίζουν. Ε, θα είμαστε πολύ πολύ αυστηροί λοιπόν. Τώρα όσον αφορά τα σύνθετα υλικά, ε, θα το δούμε γιατί ε, αν όντως ήδη συλλέγονται χωριστά, συν ε, το γεγονός ότι τα απόβλητα από οικοδομές, οικοδομικά υλικά θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά, νομίζω θα έχουμε κάτι πολύ θετικό για την κυκλική οικονομία εν γέννη. Okay. Can I suggest to make a small jump? Να κάνουμε ένα μικρό άλμα. Είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει ε, και με το τι θα συζητήσουμε συνέχεια. Αυτό είναι η πρόληψη ε, ε, παραγωγής αποβλήτων. Είναι ερώτηση 18 και 19. Αποφυγή δηλαδή καλύτερα παραγωγής. Yes, Chair. With... Με χαρά, Πρόεδρε. Έχει απόλυτη σημασία και αυτό το θέμα γιατί η ε, αποφυγή παραγωγής αποβλήτων είναι ψηλά στην ιεραρχία. Παρόλα αυτά όμως είναι σχετικά ένα νέο θέμα για τα κράτη-μέλη και νέα έννοια. Γιατί ήρθε στην οδηγία πλαίσιο το 2008 μόλις και ζητεί να εγκριθούν προγράμματα αποφυγής παραγωγής μέχρι το Δεκέμβριο του 13, δηλαδή πριν από 2,5 χρόνια, έχουν ε, εγκρίνει και εφαρμόσει ε, αυτά τα προγράμματα οι περισσότερες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει προσφύγει από παραλήψη 108 κρατών που δεν το κάνουν. Εξ αυτών τέσσερα, Σλοβενία, Κροατία, Ρουμανία και Βέλγιο, Βαλονία δηλαδή, δεν έχουν ακόμα εγκρίνει τέτοια προγράμματα. Η υποχρέωση αναθεώρηση των προγραμμάτων ε, είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουν αυτό οι οργανισμοί που παίζει ρόλο κλειδί για την πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και βελτίστων πρακτικών. Το έχει κάνει λοιπόν αυτό ο οργανισμός το 2014 και 2015 ξεολόγησε τα προγράμματα και όλα τα προγράμματα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις οδηγίας. Αλλά επειδή είναι σχετικά νέα ακόμα όλα αυτά τα προγράμματα, είναι πολύ νωρίς για να αποτιμήσουμε την αξιοπιστία, μάλλον την αποδοτικότητα. Η ε, νομοθεσία οδήγησε σε σοβαρό προβληματισμό ε, για την αποφυγή παραγωγής αποβλήτων, καλύπτει πολλούς τομείς. Τώρα απομένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί στην πράξη και πώς οι διάφορες διοικήσεις θα μπορέσουν να αλλάξουν τις νοοτροπίες. Στη νέα νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο να ενισχύσει αυτές τις ε, διατάξεις, τα κράτη-μέλη να ορίσουν και δείκτες αλλά και στόχους για τον έλεγχο αυτών όλων. Και σε σχέση με ε, την σπατάλη τροφίμων και τα απόβλητα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να το κοιτάνε και αυτό σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και μάλλον μεθοδολογία που εκπονείται αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Μποναφέ. Πολύ χαίρομαι που ακούω αυτά τα λόγια από το στόμα του κύριου Διευθυντή. Και εγώ θεωρώ ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί είναι το πρώτο βήμα στην ιεραρχία των αποβλήτων, αλλά είναι πολύ σημαντική γιατί η οπτική δεν είναι αναθεώρηση της οδηγίας για τα αποβλητά αλλά είναι η ευρύτερη οπτική της κυκλικής οικονομίας. Όταν λειτουργεί η πρόληψη σημαίνει ότι εκ των προτέρων έχουμε κάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες ε, καινοτομίας, διάφορα μοντέλα business που μας οδηγούν προς την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι στο θέμα της πρόληψης ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα, ε, καθορίζοντας και δείκτες ε, που θα πρέπει γρήγορα να μας δώσουν στοιχεία για την πρόληψη. Όμως δεν κατάλαβα καλά Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τις δράσεις που προβλέπονται για τα κράτη που μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει προσχέδια εφαρμογής. Ε, ευχαριστώ. Όκεν. Ευχαριστώ που σήμερα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Τριάντα χρόνια περιμέναμε για τις πλαστικές σακούλες. Κάπου τόσο. Και όταν πέρασε η νομοθεσία, πολλές διαμαρτυρίες, όχι από εσά, αλλά από την Κομισιόν και από το προσωπικό της Κομισιόν, ότι δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατο να το εφαρμόσουμε. Και τώρα βλέπουμε ότι τελικά λειτουργεί. Και τέλεια. Και πολύ αποτελεσματικά. Πρόσφατα ακούσαμε από την Ολλανδία, για να ενημερώσω και τον κύριο Τίμερμαν, ότι να τον ενημερώσω ήταν τεράστια επιτυχία. Τώρα και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες. Αλλά τώρα θέλουμε είναι ότι έχουμε συγκεκριμένους στόχους Πότε θα υποβάλλετε, προτείνετε παρόμοια χρήσιμα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρώτη προτεραιότητα στην ε, πρόληψη στο πλαίσιο της διαχείρισης αποβλήτων. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις? No. And then... Miss Yes. Εγώ θα ήθελα απλά να τονίσω να θέσω την, ε, την ε, εξή ερώτηση. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν έχει προσπαθήσει να κάνει διάφορα πράγματα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων στα κρατημέλη. Όμω. Όμως, ενώ Έχουμε πολλά μόνιμα ζητήματα που χρονίζουν και τα στατιστικά. Θα ήθελα να δούμε, να ελέγξουμε μια φορά τι θα κάνει τελικά η Κομισιόν. τα προβλήματα οφείλονται στην επιλεξιμότητα. Πόσο μεγάλο τμήμα είναι οι ορισμοί, οι ευθύνε και αυτό θα ήταν σημαντικό να το γνωρίζουμε. Και τέλος, εξίσου σημαντικό είναι πότε η Κομισιόν και αν η Κομισιόν θα αναλάβει νομική δράση, ε, νόμιμη δράση ε, κατά των κρατών που δεν ε, εκτελούν σωστά την ισχύουσα νομοθεσία γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε στα επόμενα βήματα όταν δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Και το μήνυμα που θα έστελνε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ότι δεν το παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα. Δεν απασχολεί. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συγκεκριμένων μέτρων για την πρόληψη δημιουργίας ε, ε απορριμμάτων. Ε, θα δείτε το άρθρο 9 της πρότασης ε, ε, πλαίσιο, οδηγίας πλαισίου. Εκεί αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα το κείμενο. Ενθάνιση της χρήσης ε, συγκεκριμένων προϊόντων που είναι ανακυκλώσιμα, επιδιορθώσιμα, επισκευάσιμα κλπ. Εντοπισμός ε, των ε, προϊόντων με, που είναι βασικές πηγές πρώτων υλών, χρήση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης, για παράδειγμα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και αποβλήτων κατά τη διαδικασία εξαγωγής ορυκτών και ως μέθοδο προτείναμε κάθε κράτος μέλος να ε, εντοπίσει τους δικούς του εταίρους ε, με τους οποίους θα συμματχίσει ε, για την μείωση, για την βελτίωση της πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων και αποβλήτων ανάλογα με τα απορρίμματα τα οποία δημιουργεί κατά κεφαλήν η συγκεκριμένη χώρα. Κυρία είναι. Ε, προσπάθησα να απαντήσω στην αρχή, στην εισαγωγική μου παρέμβαση σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι πρέπει να το επαναλάβω. Ε, πρόκειται για οδηγίες οι οποίες πρέπει να μεταγράφονται ορθά και να εφαρμόζονται. Ε, η ίδια νομοθεσία δεν είναι τόσο περίπλοκη. Δίνει μια κατεύθυνση, σαφή κατεύθυνση όμως. Υπάρχουν πάντοτε δυνατότητες νο, νόμιμων εκθέσεων για πράγματα που δεν συμβαίνουν. Δηλαδή υπάρχουν παραθυράκια που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να δηλώνουν ότι έχουν ανακυκλώσει κάτι το οποίο δεν έχει στην πραγματικότητα ανακυκλωθεί, έχει υποστεί ταφή ή καύση για παράδειγμα. Ελπίζω ότι η έκθεση η οποία θα είναι διαθέσιμη νομίζω ελπίζω αυτή τη βδομάδα από τη Σιμώνα Μποναφέ θα σχολιάσει αυτό το θέμα και θα προτείνει αυτά που προτείνουμε κι εμείς Πρόεδρος, ωραία ας περάσουμε στην τελευταία ομάδα ερωτήσεων ε, καθορισμός, ε, μάλλον υπολογισμός στόχων ερωτήσεις 13 και 14 Μπορώ να ζητήσω από την Κομισιόν να απαντήσει. Um, um, Η φυστάμενη νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να, ε, να χρησιμοποιούν μία από τις τέσσερις υπάρχουσες μεθόδους υπολογισμού και αυτό είναι και το θέμα το οποίο σχολέζαμε και προηγουμένως. Αυτό επιτρέπει τον ορισμό του, του των ε, δημοτικών αποβλήτων ε, για το τι μετράμε και πού το μετράμε. Σε ό,τι αφορά το τι είναι ε, δημοτικά απόβλητα, τα κράτη-μέλη μπορούν να μετρήσουν είτε το συνολικό, ε, ε τη συνολική ροή, ε, μόνο κάποια τμήματα, τα, πολυ, τα των οικοκυριών ή νοικοκυριών και δημόσιων υπηρεσιών. Τώρα το πού μετρώνται τα απορρίμματα και πάλι έχουμε διάφορες μεθόδους. Πρώτον, στο σημείο διαλογής ή συλλογής, αν δεν υπάρχουν σημαντικές απώλειες, ή στην είσοδο των αεροστάσεων εκκύκλωσης. Τώρα, τι σημαίνει σημαντικέ απώλειε. Δεν το καθορίζει ο νόμο, οπότε τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε από τι μεθόδου και μα λένε, κάποια κράτη-μέλη μα ε, λένε ότι εφαρμόζουν το 0% με την τάδε μέθοδο, άλλοι μα λένε 30%. Το... Ε, οπότε στην πραγματικότητα δεν μετράμε ακριβώ το τι πραγματικά να κυκλώνεται και αυτό προφανώς πλήττει την αξιοπιστία των δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν προτείνει ένα κοινό ορισμό των δημοτικών ε, απορριμμάτων και πιο κοινού κανόνες για την μέτρηση. Ο κοινό ορισμός που προτείνουμε προέρχεται από την Eurostat και από τον ορισμό της Eurostat και του ΟΣΑ τον οποίο χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη εδώ και καιρό ε, χρησιμοποιούσαν μάλλον ε, όταν ανέφεραν στο γύρο στα τα στοιχεία τους σε εθελοντική βάση. Είναι η πιο ακριβής μέθοδος. Σε ό,τι δεν αφορά το πού γίνεται η μέτρηση, προτείνουμε να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι κανόνες. στα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να αναφέρουν απορρίμματα τα οποία έχουν συλλεχθεί ως ανακυκλώσιμα. Θα πρέπει να αναφέρουν και να μετρούν μόνο όσα απορρίμματα μπαίνουν στην ε, ανακύκλωση ε, ή αυτό που βγαίνει από τη διαλογή υπό την προϋπόθεση όμως ότι ε, η απώλεια μέχρι να μπουν στην ανακύκλωση είναι κάτω από 10% και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά που μπαίνουν στην ανακύκλωση πραγματικά ανακυκλώνονται. Το, η, ο όρος μη σημαντικές απώλειες ε, θα πρέπει να γίνει πιο σαφής. Ε, πρόκειται για υλικά τα οποία βρίσκονται στα απορρίμματα ακόμα και μετά τη διαλογή αλλά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν κλπ. Γνωρίζουμε ότι για τα, τις βασικές κατηγορίες απορριμμάτων ε, η ανακύκλωση απαιτεί να είναι πολύ πιο ποιοτική η διαλογή. Ε, το σημαντικό είναι να βρούμε την πιο καλή λύση έτσι ώστε πραγματικά να μετράμε το τι ανακυκλώνεται αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να μας εννοούν και για το πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα αυτών των στοιχείων. Εμείς έχουμε λάβει υπόψη το επίπεδο απόδοση κάθε κράτο μέλο και τις διαφορές στην, ε, στον υπολογισμό των δημοτικών απορριμμάτων. Έχουμε αναπτύξει ένα πραγματικά περίπλοκο μοντέλο ε, ε, για, την, για τον υπολογισμό των απορριμμάτων και λαμβάνουμε υπόψη το input κάθε κράτους μέλους ε, και τα διάφορα, τις διαφορετικές μεθόδους για τον τόπο υπολογισμού. Γνωρίζουμε την κατάσταση, δηλαδή, την έχουμε λάβει υπόψη. Την, η αξιολόγηση που κάνουμε έλαβε υπόψη τις σημερινές αποδόσεις και τα μελλοντικά σχέδια καθώς επίσης και τη σύνθεση και διαχείριση των αποβλήτων σε κάθε χώρα. Επίσης, ζητήσαμε από τις αρχές να μας επιβεβαιώσουν ορισμένα στοιχεία. Αυτό θα μας δώσει επαρκείς λεπτομέρειες για να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία μεταξύ των κρατών μελών. Ταυτόχρονα θα καταφέρουμε αυτόν τον τρόπο να βεβαιωθούμε ότι οι στόχοι που προτείνουμε είναι ρεαλιστικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όκεν. Μια σύντομη ερώτηση. Θέλω να ξέρω αν προβήκατε σε κάποιες ενέργειες, αν κάνατε κάτι, για να εξασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη τηρούν τη τρέχουσα νομοθεσία και επίσης τι κάνει την Κομισιόν να πιστεύει ότι το 10% θα βελτιώσει την εφαρμογή. Τι κάνατε στην πράξη για να λειτουργήσει. Και σεβαστήκατε αυτό το 10% στην εφαρμογή. No, please. Um... Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω το 5% από που βρέθηκε στο νόμο. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Αυτό που ισχύει τώρα και αυτό που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Έχουμε μελιτές απώλειες. Αλλά το κράτος κάθε μέλος ε, το ερμηνεύει κατά το δοκούν και ορισμένα κατά χρόνια κιόλας. Και φτάνουμε μέχρι το 30%. Αυτό θέλουμε να κλείσει το παραθυράκι, να πούμε έναν αριθμό που να είναι ρεαλιστικός και να βασίζεται στα όσα γνωρίζουμε και τι συμβαίνουν στην πραγματικότητα, στα κέντρα διαλογής των αστικών αποβλήτων. Αυτό μπορεί να γίνει και από εκεί και πέρα αυτό πάντα θα πρέπει να είναι εξαίρεση. Ο κανόνας να είναι να μας ε, δηλώνουν ε, στην τελική ανακύκλωση την μπαίνει. Αυτό το 10% θα ισχύει μόνο κάτι εξαίρεση και μόνο υπό την προπόθεση ότι τα κράτη-μέλη ε, εξηγούν τη μεθοδολογία και πώς τα μετρούν όλα αυτά. Και αν δεν είμαστε πεπισμένοι ότι είναι γερή, στιβαρή και αξιόπιστη μέτρηση, δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Τώρα έτσι είναι κάτι γενικό, χωρίς κανένα μετρήσιμο στοιχείο. Με το 10% πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε αρκετά υψηλή ποιότητα της ροής στην ανακύκλωση. Και για το γυαλί, ας πούμε, ε, και το 10% πολύ είναι. Και δεν ε, το αξιοποιούν αρκετά τα κρατημέλη. Το ξέρουν και τα κρατημέλη και οι ανακυκλωτές και οι πελάτες των ανακυκλωτών που το αγοράζουν και τα χρησιμοποιούν στη συνέχεια η κλάδη αυτή της οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, προτείνω να κλείσουμε εδώ αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή της οδηγίας ε, πλαίσιο για τα απόβλητα και τις συσκευασίες. Ευχαριστούμε την ε, Κομισιόν. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις μπορούμε να συνεχίσουμε για τη συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση. Και εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Θέλω μόνο να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση Τη Επιτροπή Περιβάλλοντο θα είναι στι 15 και 16 Ιουνίου εδώ στι Βρυξέλλε. Σα ευχαριστώ όλου. Χαίρετε.